Στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης δεν έχουμε πια την απαλλαγή του 2007 διότι αποφασίσαμε την αναβολή της. Ε, περνάμε στο σημείο 2, προϋπολογισμός 2010, τμήμα 3, Επιτροπή. Έχουμε την ε, έκθεση του Αντιπροέδρου, του κυρίου Οντή, στον οποίο θα δώσω το λόγο αμέσως. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω σχόλια να σας κάνω. Να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για τη βοήθειά της, όπως και όλους τους συναδέλφους, ε, για τις τροπολογίες που ε, παρουσίασαν στην εκθεσή μου. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω. Έχετε τα έγγραφα και μπορούμε να περάσουμε απευθείας στην ψηφοφορία. Ναι, σας ευχαριστώ. Ωραία. Να περάσουμε indica eh, eh, Να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Αν συμφωνείτε, θα κάνουμε το εξή. Θα ψηφίσουμε διανάταση ισχυρό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Συμφωνείτε? Ωραία. Λοιπόν, τροπολογία υπαριθμών 1. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Undici. Undici. Undici. Okay. Quindi eh, Εγκρίνεται η τροπολογία. Κατά. Siamo e Αποχές. Quindi Quindi emendamento... Eh. Επομένως, εγκρίνεται η τροπολογία. Να περάσουμε τώρα στην... Ε, παρακαλώ. Θέλετε να ελέγξετε ηλεκτρονικός. Ωραία. Un attimo, un attimo.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 Πέραση ψηφοφορίας. Έχετε ψηφίσει όλοι. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, Επτά υπέρ, 9 κατά και μία αποχή. Επομένως είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα από αυτό που είχαμε πριν. Απορρίπτεται η τροφοπολογία. Μήπως δεν ψήφισαν όλοι, ε, χρησιμοποιήσετε όλες τις κάρτες σας. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία, προχωράμε. Επειδή έχουμε βάλει όλοι τις κάρτες μας, για να μην έχουμε αμφισβητήσεις, θα κάνουμε όλη την ψηφοφορία ηλεκτρονικώς. Να περάσουμε λοιπόν στην τροπολογία υπαριθμών 2. Τροπολογία υπαριθμών 2, άρχεται η ψηφοφορία. Number. Απορρίπτεται η τροπολογία 12 κατά, 10 υπέρ και μία αποχή. Τροπολογία Τέσσερα. κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 23 υπέρ, κανένα κατά, καμία αποχή. Περνάμε στο δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 4, άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 12 κατά, 11 υπέρ, καμία αποχή. compatibili insieme. No, l'uno dopo l'altro. Prima il Cioè. Passiamo alla votazione. Να ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία παριθμών 3. Άρχεται η ψηφοφορία. L'emendamento è approvato con Εγκρίνεται 21 υπέρ, ένα σκατά και καμία εποχή. Περνάμε τώρα στην ε, τροπολογία 5, άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 22 υπέρ, καμία αποχή, 2 κατά. Τροπολογία υπερθμών 6. Άρχιτη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 22 υπέρ, 1 κατά, καμία αποχή. Τροπολογία. Η τροπολογία 7 καταπίπτει και περνάμε στην τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 15 ψήφοι κατά, 8 υπέρ, καμία αποχή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 9. Emendamento approvato. Εγκρίνεται η τροπολογία 22 υπέρ, 23 ε, συγγνώμη, υπέρ, Ένα κατά καμία εποχή. Τροπολογία 10. Παρακαλώ. Δεν ε, δουλεύει η κάρτα μου. Μπορεί κάποιος να διορθώσει την κάρτα του συναδέλφου. Μισό λεπτό παρακαλώ, περιμένετε.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 Πέρα της ε, τροπολογίας 10 ε, απορρίπτεται 10 υπέρ 12 κατά καμία εποχή. Περνάμε στην τροπολογία 11. Παρακαλώ. Στην τροπολογία υπαριθμών 11 η ομάδα μου πρότεινε μια προφορική τροπολογία. Θα σας τη διαβάσω και σας προτείνω να την ψηφίσουμε. Και συνεχεία έχουμε την τροπολογία της Αγιάλα Σέντερ. Αυτή η προφορική τροπολογία τι λέει, να προσθέσουμε στην παράγραφο 8. Θεωρεί ότι όλα αυτά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα έγγραφα της ε, Ένωσης που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία είναι όσο να τον πιο προσπελάσιμα από το κοινό σε κάθε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε να το ψηφίσουμε αυτό πριν από την τροπολογία 11. Αυτό προτείνω. Προτείνω πρώτα να ψηφίσουμε την προχωρική τροπολογία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και την τροπολογία για άλλα σέντερ. Μπορούμε, αλλά εμάς μας φαίνεται λίγο υπερβολικά περιοριστική η τροπολογία για Λασέντερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Γιάλα Σέντερ. Με συγχωρείτε επειδή τα γαλλικά μου δεν είναι πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να ζητήσω τι σημαίνει relevant de la legislation στα γαλλικά. Σημαίνει μόνο τη νομοθεσία ή μπορεί να σημαίνει και όλα τα προ ε, παρασκευαστικά ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι κάτι πιο ευρύ από την νομοθεσία, διότι αυτό που θέλουμε είναι να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλες τις γλώσσες. Ε, εγώ συμφωνώ υπό την προϋπόθεση ότι το relevant legislation δεν σημαίνει αποκλειστικά και μόνο την νομοθεσία, αλλά μπορεί να σημαίνει και κάποια προπαρασκευαστικά έγγραφα, κάποια ανακοίνωση, ε, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας δίνουν συνήθως. Συμφωνώ δεν, ήθελα, δεν είχα πρόθεση να είναι όλα εννοείται, διότι έχουμε και οικονομικά προβλήματα επί του παρόντος, αλλά θα ήθελα τουλάχιστον να μην αφορά αποκλειστικά και μόνο την νομοθεσία, διότι κάποιες φορές υπάρχουν συστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι πολύ πιο ε, ε χρήσιμες για τους πολίτες από την ίδια την νομοθεσία, διότι όλοι οι πολίτες δεν είναι νομικοί, δεν είναι τα παραρτήματα. Ξέρω ότι η κυρία Γκρέσλερ έχει αιμονή με τα παραρτήματα που δεν θα μεταφραστούν. Εμένα δεν με πειράζει να μην τα μεταφράσετε, θα προτιμούσα να τα μεταφράσουμε, αλλά ε, δεν μιλάμε όλοι αγγλικά και θέλω τα υπόλοιπα. Ε, ζητώ συγγνώμη που τώρα ενώ ψηφίζουμε θα κάνουμε αναγκαστικά μια πολιτική ανταλλαγή απόψεων. Ακόμα και όταν είναι μόνο στα αγγλικά τα παρατήματα είναι πολύ σημαντικό να τα κρατήσουμε γιατί είναι πολύτιμα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε ότι αυτό που αφορά την νομοθεσία, το relevant de la législation, μπορεί να περιορίσει το εύρος των μεταφράσεων. Αν τώρα ε, αποσύρετε δική σα τροπολογία, να βάλουμε που άπτεται των κοινοβουλευτικών εργασιών. Επομένω, αυτό σημαίνει όλε οι εργασίε του Κοινοβουλίου. Όχι μόνο νομοθεσία, έτσι, αλλά και τα πάντα όλα, και τα υπόλοιπα πράγματα και τα νομοθετικά κείμενα και τα υπόλοιπα. Από ό,τι κατάλαβα, αποσύρετε τη δική σας τροπολογία βάσει των όσων και είπε σήμερα ο κύριος, ε, τώρα συγγνώμη, ο κύριος Οντή. Επομένως ψηφίζουμε την ε, προφορική τροπολογία που παρουσίασε ο κύριος Οντή. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 24 υπέρ, κανένα κατά, καμία αποχή. Η τροπολογία 11 λοιπόν αποσύρεται και περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 12. Άρχεται η ψηφοφορία. 23. Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ, κανέν, καμία κατά, μία αποχή. Τροπολογία περισμών 13, άρχεται η ψηφοφορία. Εμενταμέντο Απορρίπτεται. 8 υπέρ, 17 κατά. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 25 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, καμία εποχή. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, η τροπολογία 15. Votazione aperta. Emendamento approvato. Εγκρίνεται. 25 ψήφοι υπέρ, κανένα κατά, καμία εποχή. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Emendamento respinto con 16 voti, 8. 8 υπέρ, 16 κατά, μία αποχή απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 17, άρχιτη ψηφοφορία. Emendamento respinto con 17. Απορρίπτεται. 8 υπέρ, 17 κατά. Να περάσουμε τώρα ο κύριο Σοντή, παρακαλώ. Με μικρόφωνο, κατά προτίμηση. Για την παράγραφο 12. Θα ήθελα να κάνω πάλι μια προφορική τροπολογία. Σήμερα το πρωί τη σκέφτηκα. Είναι για την τακτοποίηση αυτών που οφείλουν τα κράτη-μέλη για τις συντάξεις των, των μελών του προσωπικού της Ένωσης. Τη στιγμή που δούλεψα αυτό το σχέδιο έκθεσης, δεν είχα δει τους ετήσιους λογαριασμούς. Ε, κανονικά το νούμερο είναι 36,9 δισεκατομμύρια 31 Δεκεμβρίου του 2008. Να πούμε, που εκτιμόταν 36,9 ε, δισεκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Τελικά αυτό αφορά την τροπολογία 11, διορθώνει ο μιλητής, όχι 12. Τα νούμερα αυτά του 2008 βγήκαν στο πρώτο εξάμεινο του 2009. Να πούμε ότι εκτιμάται σε 36,9 δισεκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Να διορθώσουμε αυτό το νούμερο. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Επιτρέψτε μου, επειδή απλά είναι επικαιροποίηση ενός ε, στοιχείου που απλά δεν ήξερε ο εισηγητή, ε, νομίζω ότι μπορούμε να το δεχτούμε χωρίς να χρειάζεται να ξαναψηφίσουμε μια παράγραφο την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Είναι μια τεχνική διόρθωση την οποία μπορεί να επικαιροποιήσει η Γραμματεία με βάση τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ κι εγώ, μια απλή διόρθωση είναι, δεν υπάρχει λόγος να ψηφίσουμε, συμφωνούμε.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 26 Εγκρίνεται 26 ψήφοι υπέρ, καμία αποχή, κανένα κατά. Περνάμε τώρα στην τροπολογία υπερθμών 19, άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 7 υπέρ, 18 κατά, μία αποχή. Τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 22 υπέρ 3 κατά μία αποχή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Emendamento approvato con 23 voti favorevoli. Εγκρίνεται 23 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Emendamento approvato con 23. Εγκρίνεται 26 υπέρ, καμία αποχή, κανένας κατά. Τροπολογία υπέρ 23, άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 10 υπέρ, 15 κατά, μία αποχή. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με τις τροπολογίες. Να ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του κειμένου, άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 25 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ντί, τον Αντιπρόεδρο για τη δουλειά του και να προχωρήσουμε στην, ε, στην υπόλοιπη μερίσια διάταξη. Eh, Να περάσουμε τώρα σε μία σύντομη περίληψη, διότι λάβατε όλοι και το σχετικό έγγραφο ε, για τη συνεδρίαση των συντονιστών που έγινε χθες το απόγευμα μετά από την συνεδρία της Επιτροπής μας. Ορίσαμε τους εισηγητές για τα θέματα που μας απασχολούν επί του παρόντος. Μπορείτε να τα δείτε αυτά στο σημείωμα το οποίο μας διαβιβάστηκε από τη Γραμματεία. Το ίδιο αφορά και στους ε, εισηγητές για την απαλλαγή για το 2008, καθώς επίσης και τις αποφάσεις ε, για την αναστολή των ε, θεμάτων που είχαν αναβληθεί από το Μάρτιο του 2009 Έχουμε και τις ε, γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίες και το σημείο 5, την ειδική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορείτε να βρείτε όλες τις ε, ομάδες που συμμετέχουν ε, για τα κείμενα, τη σύνταξη αυτών των κειμένων. Έπρεπε επίσης να αποφασίσουμε και για κάποια θέματα που αφορούσαν στις αντιπροσωπίες, τις ακροάσεις και τις μελέτες ε, οι οποίες πρέπει να προβλεφθούν για τους επόμενους μήνες, κυρίως όσον αφορά στις αντιπροσωπείες και τις ακροάσεις, ε, το θέμα ήταν ιδιαίτερα επίγον, διότι όπως μας είχε υποδείξει και η Γραμματεία, πρέπει να αποφασίσουμε μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Θα βρείτε λοιπόν στο κείμενο κάποιες μελέτες οι οποίες προτάθηκαν και εγκρίθηκαν εχθές, αλλά έγινε και η συζήτηση για κάποιες ακροάσεις, τις οποίες θα δείτε στο Β2. Για τις αντιπροσωπείες έχουν υποδεχθεί οι εξής χώρες, η Ιταλία ε, για τη Λομβαρδία, το Αμπρούτσο, την Καλάβρια και την Κατάνια, ε, Βουλγαρία, Κωσυφοπέδιο, Ελλάδα, Κύπρος και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Όπως μου είπε η γραμματεία, ο κύριος Μπράουν σήμερα το πρωί, Από αυτές τις αντιπροσωπείες, κατά πάσα πιθανότητα, μόνο τρεις θα μπορέσουμε να κάνουμε μόνο μέσα στο 2010 και οι υπόλοιπες θα πρέπει να μεταφερθούν στο 2011. Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο λύσεις. Ή θα αποφασίσουμε τώρα ποιες από τις τρεις ε, αποστολές θέλουμε να κάνουμε το 2010 ή θα το αναβάλουμε για μια επόμενη συνεδρίαση των πολιτικών ομάδων με τη Γραμματεία και μεταξύ των χωρών αυτών θα επιλέξουμε ποιε θα πρέπει να γίνουν πρώτα εντό του 2010. Αν θέλετε να το σκεφτείτε λίγο, μπορεί να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω και να δούμε. Αλλιώ μπορούμε να αποφασίσουμε και τώρα αν βρούμε ποιε ε, είναι οι τρει βασικέ ομάδε Από τι χθεσινέ ενδείξει. κατάλαβα ότι το ΕΛΚ, ε, ο κύριο Γκράσου είχε υποδείξει την ε, Ουγγαρία. Ο κύριος Γκέγερ ήθελε να πάμε στην Ελλάδα, αν δεν θυμάμαι καλά, και οι φιλελεύθεροι ήθελαν να πάμε στην Ιταλία. Επομένως, ή αποφασίζουμε έτσι ή μπορούμε να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα και να το παραπέμψουμε στη γραμματεία ε, και τις πολιτικές ομάδες την επόμενη εβδομάδα. Αλλά η προθεσμία είναι 7 του μηνός, οπότε σε λίγες μέρες πρέπει να έχουμε αποφασίσει. Παρακαλώ. Ο κύριος... Θέλω να ρωτήσω εάν κατάλαβα καλά την πρότασή σας. Εάν δεν αποφασίσουμε σήμερα, ή επειδή πρέπει να αποφασίσουμε μέχρι τις 7 Δεκάτου, τι θα κάνουμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σας το είπα. Μπορούμε να αποφασίσουμε σε μια συνεδρίαση της γραμματείας με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Να δούμε σε ποιο από τα τρία κράτη θα δώσουμε προτεραιότητα. Τις ε, επόμενες μέρες θα κάνουμε αυτή τη συνεδρία, μέχρι τις 7 του μηνός. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Έχουμε τρεις προτάσεις από τρεις ομάδες. Ουγγαρία, Άλντα, Ιταλία και η S&D επίσης. Τρεις ομάδες λοιπόν τρεις οψιών. Μπορούμε να αποφασίσουμε σήμερα αν θέλετε. Εάν ορισμένες ομάδες δεν είναι έτοιμες να αποφασίσουν μπορούμε να το αναβάλουμε. Αλλά έχουμε τρεις προτάσεις ε, από χτες και οι τρεις είναι αποδεκτές. Γιατί να μην πάρουμε αυτές τις τρεις και να επιλέξουμε. Μετά από αυτά που μου είπε η γραμματεία, Καλύτερα θα ήταν βέβαια να αποφασίσουμε σήμερα, αν μπορούμε. Όσο νωρίτερα αποφασίσουμε, το καλύτερο. Αλλά εγώ σα δώσω και μια εναλλακτική λύση, έτσι, για να είμαστε πιο άνετοι. Ο κύριο Σοντή. Μία προσωπική γνώμη να εκφράσω για την Κροατία. Γιατί αν αύριο οι, Ιρλανδοί έχουν την εξυπνάδα να υπερψηφίσουν τη Λισαβόνα, ε, τότε οι τροποποίησεις ε, που συμφωνήσαμε με τον Επίτροπο θα μπουν στην ε, Συμφωνία Ένταξης Κροατίας και θα επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία. Όπως κάναμε και στο Κοσφοπέδιο ε, στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία, λοιπόν, δεν θα ήταν καλό να πάμε τώρα στην Κροατία για να είμαστε έτοιμοι για αυτή την πολιτική επιτάχυνση. Ξε... Και εξάλλου, η διαπραγμάτευση των συνόρων ε, Σλοβενίας, Κροατίας ε, επιταχύνεται και αυτή. Όλα πηγαίνουν καλά. Επομένως, τα πράγματα για την Κροατία επιταχύνονται. Αυτή είναι μια προσωπική μου γνώμη. Τι λέτε, ο κύριος Λιμπεράσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέποντας αυτές τις τρεις χώρες που προτείνονται, θέλω να σας θυμίσω, πέρσι επισκεφθήκαμε τη Βουλγαρία, δεν ξέρω εάν πρέπει κάθε χρόνο να πηγαίνουμε ή κάθε δεύτερο χρόνο. Είχα τότε την έγκρισή σας να συμμετάσχω στην αποστολή της Βουλγαρίας. Φέτος νομίζω δεν χρειάζεται. Ο κύριος Τσαρνέσκι. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω την πρότασή σας για την Κροατία δέχομαι. Πιστεύω βέβαια ότι η έγκριση, η απόρριψη της Λισαβόνας δεν θα επηρεάσει την ένταξη ή όχι της Κροατίας, διότι θα γίνει δεκτή η, έγκριση, η ένταξη της Κροατίας, οπότε θα γίνει η ενταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι η επίσκεψη στη χώρα αυτή είναι σημαντική και υποστηρίζω την πρότασή σας για την Κροατία, ιδίως επειδή δεν νομίζω ότι είχαν και πολλά προβλήματα με την προενταξιακή ενίσχυση που τους δόθηκε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γκέιγε, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλα τα κράτη που ανέφερα προηγουμένως, ε, για αυτά έχει προβλεφθεί μία επίσκεψη. Το θέμα είναι να δούμε ποια είναι η προτεραιότητα. Μέχρι το 2010 θα κάνουμε τρεις ή τέσσερις τέτοιες αποστολές και οι υπόλοιπε το 2011. Το θέμα είναι να δούμε τις προτεραιότητες τώρα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και άλλες επισκέψεις. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω την πρόταση του συναδέλφου Οντί και προτείνω του χρόνου να εγκρίνουμε την αποστολή στην Κροατία ε, ε, βεβαίως υποστηρίζω, μου αρέσει και η ιδέα της Ελλάδος και της Ιταλίας, ιδιαίτερα με την ενίσχυση που δόθηκε μετά τη μεγάλη καταστροφή στην περιοχή του Αμπρούτσο, ε, μπορούμε να πούμε Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία με αυτή τη σειρά και να, να κάνουμε αυτό τον κατάλογο προτεραιότητας. Κροατία, ε, Ελλάδα, Ιταλία. Mm, θα δώσω το λόγο μια στιγμή στο ΕΛΚ. Γιατί επειδή χθε η κυρία Γκρέσλε είχε μιλήσει, μιλήσει και για την Ουγγαρία, θα μπορούσαμε να κάνουμε Ιταλία, Κροατία που την ήθελε και η κυρία Γκρέσλε και Ελλάδα. Την ε, Ιταλία, Κροατία και Ελλάδα το 2010 και όλες τις υπόλοιπες να τις αφήσουμε το 2011, όπως στην Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Η Ουγγαρία Ιταλία, Ελλάδα και μετά Κροατία. Γιατί χτες λίγο πολύ είχαμε συμφωνήσει. Το 2007 έγινε αποστολή στην Ελλάδα. Ιταλία, Ουγγαρία και Ελλάδα νομίζω. Και μετά τέταρτη στη σειρά η Κροατία η Κροατία. Ε, Ουγγαρία, Ιταλία, Ελλάδα, τέταρτη Κροατία. Αν θέλετε να κρατήσουμε τότε την Ουγγαρία, θα πρέπει να κάνουμε Ουγγαρία, Ιταλία, Κροατία. Και να βάλουμε τότε την Ελλάδα για το 2011. Λοιπόν, ε, φαίνεται σαν να παίρνουμε μία απόφαση για το πού θα πάμε τις επόμενες διακοπές. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή του συστήματος ελέγχου. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Και γι' αυτό υποστήριξα και την κυρία Γκρέσλα χτες. Ότι πρόκειται εδώ για την ε, έλεγχο του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, τον οποίο έχουμε προγραμματίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα, από πολιτικής απόψεως, πού πέφτει το κέντρο βάρους και ε, ποια είναι, ποια είναι η πιο σημαντική πολιτική πτυχή, ας πούμε, για την απόφαση μας πρέπει να ακολουθεί τη βασική προτεραιότητα που είναι η σωστή εφαρμογή του ελέγχου. Πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα και με σοβαρότητα και να προχωρήσει το θέμα του ελέγχου στην Ελλάδα. Γι' αυτό εμένω στην αποστολή στην Ελλάδα το 2010. Πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφο, Νομίζω ότι να περάσουμε στις τέσσερις από το στολές. Ιταλία, Ουγγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Ε, να κάνουμε αυτές τις τέσσερις λοιπόν στο 2010 και τις υπόλοιπες αποστολές το 2011. Και αν συμφωνείτε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Για λόγους πολιτικής ισότητας θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ένα παλαιό κράτος μέλος, Ελλάδα και η Ιταλία και ένα νέο κράτος μέλος, Ουγγαρία π.χ. Και μια χώρα που ε, θα ενταχθεί, Κροατία, παλιά, νέα, μέλουσα. Το ίδιο λέμε. Η, προτεραιότητα του 2010 είναι Ιταλία, Ουγγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Και στις υπόλοιπες ε, χώρες που αναφέραμε χθες θα πάμε το 2011. Συμφωνούμε? Έχουμε λίγο χρόνο. Αν κάποιος θέλει να μιλήσει για τις μελέτες, ενώ γιατί για τις, ακροατι... ακροάσεις και τις αποστολές. Είχαμε την αποστολή της 7 Οκτωβρίου. Για τις μελέτες έχουμε περισσότερη προθεσμία. Αν λοιπόν κάποιος βουλευτής θέλει να προτείνει κάποια μελέτη την επόμενη φορά, στην επόμενη συνεδρίαση, να το προτείνουμε. Ο κύριος Λιμπεράσκη. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Θέλω να επανέλθω στο θέμα των αποστολών, γιατί έγινε η πρόταση να διαλέξουμε μια, ένα παλιό κράτος μέλος, καινούριο και μελλοντικό. Πολωνία, Ουγγαρία είναι νέα κράτη-μέλη και εάν μας ανησυχούν διάφορα, διάφορες καταστάσεις όπως την Ελλάδα, προτείνω την εξής σειρά. Η Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία τέταρτο η αποστολή, τέταρτη θέση αλλά να βάλουμε τις προτεραιότητές μας εκεί που χρειάζεται, εκεί που υπάρχει ανάγκη και όχι βάσει παλαιών ή νέων κρατών μελών και πολιτικών αποφάσεων. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε μετά. Φυσικά δεν πρόκειται για αντιπροσωπείες που θα πάνε να κάνουν αποστολε, ε, διακοπές, αλλά θα ελέγξουν κάποιες κατατά, καταστάσεις. Γι' αυτό εντοπίσαμε και αυτές τις συγκεκριμένες χώρες, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος ως Επιτροπή να πάμε. Αλλά δεν θα αποφασίσουμε σήμερα το πώς ε, θα διεξαχθούν αυτές οι αποστολές. Αυτό το κάνουμε άνετα τις επόμενες ημέρες. Η κυρία Γέλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το θέμα των ε, μελετών. Απλά σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να κάνουμε νέες προτάσεις. Αλλά για τον κατάλογο που έχετε ήδη, που υποθέτω ότι είναι αυτός που συμφώνησαν οι συντονιστές, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στις δύο μελέτες που αφορούν στις ε, δημοσιονομικές προοπτικές, δηλαδή την εφαρμογή των διαφορετικών υγειοργικών ταμείων για το 2007-2013. Εχθές είδαμε ότι αυτό που είχαμε και στο 2000-2007 ήταν πάρα πολύ νωρίς για να καταλήξουμε στα, σε συμπεράσματα ε, και αυτό ε, ισχύει και τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα και σε οριστικές συστάσεις οι οποίες ε, ε, απλά μια ενδιάμεση τοποθέτηση θα ήταν. Ενώ για το 2094 έως το 2000 έχουμε μείνει πεινασμένοι και η Κομισιόν μας έδωσε κάποια στοιχεία και η όλα εχθές μας έδωσε κάποια στοιχεία για παρατυπίες. Επομένως θα θέλαμε, εάν υπάρχουν κάποιες μελέτες που έχουν γίνει, εγώ δεν λέω τίποτα γιατί δεν τις γνωρίζω και δεν τις ε, έχω δει. Έχω δει κάποια στοιχεία που μας έδωσαν άλλα θεσμικά όργανα, αλλά θα ήθελα τουλάχιστον να μπορέσουμε να εξετάσουμε για να έχουμε και μια εικόνα του τι ακριβώς έγινε, να έχουμε μια συνέχεια. Τι έγινε το 1994-2000, 2000-2007 και να είμαστε προετοιμασμένοι για του χρόνου που θα γίνει μια ενδιάμεση εξέταση για να δούμε και πώς έχουμε προοδεύσει και να έχουμε και οριστικά αποτελέσματα. Να λέμε απλά ότι έχουμε ποικίλα αποτελέσματα και τι γίνεται με τα διαρθρωτικά ταμεία, ε, ξέρετε ότι δεν μας δίνει στοιχεία τα πράγματα τα οποία έχουν ε, σχεδόν ε, ολοκληρωθεί, διότι υπάρχουν πράγματα που είναι ανοιχτά και για το 1994 1999 Να δούμε λοιπόν τι ξέρουμε για αυτά, τι ξέρουμε για το 2000-2006 και να δούμε και τι γίνεται με τις ε, παρούσες προοπτικές, γιατί είναι συνοχιζόμενες και θα μπορέσουμε να βγάλουμε και κάποια σχετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Όπως είπα προηγουμένως, έχουμε χρόνο για να κάνουμε όλες αυτές τις προτάσεις. Εσείς λοιπόν έχετε χρόνο για να δείτε τι πρόταση θα κάνετε που θα και θα την υποβάλλετε στην Επιτροπή και στις ομάδες. Το επόμενο σημείο, το σημείο Γ, πρόκειται για τις ακροάσεις των Επιτρόπων. Αρχικά είχαμε σκεφτεί τη δυνατότητα οι ακροάσεις ήταν πάρα πολλέ και είχαμε <laughs> λίγες συνεδριά στη διάθεσή μας. Επομένως, έγινε μια πρόταση από τον εισηγητή, τον κύριο Λιμπεράσκη, να μειώσουμε τον αριθμό των ακροάσεων. Από τη συζήτηση που είχα χθες με τους συντονιστές προέκυψε η ανάγκη να ακούσουμε όλους τους επιτρόπους. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Ε, απόλυτα σημαντικό για την Επιτροπή. Επομένω, η Γραμματεία θα πρέπει να βρει και τι μέρε και τι ώρε και τι αίθουσε για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλου του επιτρόπου. Εν συνεχεία. Αναφέρεται η συνάντηση με το Ελεκτικό συνέδριο στις 10 Νοέμβριο. Φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση με μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, βρήκαμε αυτά τα ωράρια με μεγάλη δυσκολία. Σας παρακαλώ, θέλω να έρθετε όλοι για να ακούσουμε πρώτα την ε, έκθεση και συνεχεία να γίνει συζήτηση. Γιατί, όπως είπαμε και χθε, το ελεγκτικό συνέδριο θα χρειαστεί όλο αυτό το χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είδαμε και χθε να συζητάμε, είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε όλα τα θέματα που άπτονται τη Όλαφ, και του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα πρέπει να είσαστε όλοι εδώ, ούτως ώστε να κάνετε ερωτήσεις και να ακούσετε βεβαίως ε, τις απαντήσεις. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη στο Λουξεμβούργο, ε, το απόγευμα στις 4 Νοεμβρίου θα επισκεφθούμε το Λουξεμβούργο. Ε, κατόπιν προσκλήσεως ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους του που είναι εδώ παρόντες σήμερα. Θα δούμε λοιπόν Την αναβολή για την ψηφοφορία την αποφασίσαμε και έπειτα την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης, εκθέσεως του Ελεκτικού Συνεδρίου θα την κάνουμε αυτή στις 9 Νοεμβρίου. Πάμε στο σημείο 14 της σημερινής διάταξης, την ειδική έκθεση 2-2009 Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Υγεία 2003 έως 2007, ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κύριος Φιέλνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ήθελα να διακόψω, αλλά στην πρόταση να υπάρχει ένας εκπρόσωπος ε, που μου φαίνεται τέλεια της, Ευρωπαϊ... της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, θα ήθελα η Γραμματεία να βρει έναν τρόπο με τον οποίο αυτός ο εκπρόσωπος θα, θα μπορεί να ε, αναφέρει εδώ στην Επιτροπή μας. Διότι ε, εγώ συνήθως ενδιαφέρομαι για κάποια θέματα. Θα έπρεπε ίσως να έχουμε μια ενημέρωση από καιρούς καιρούν για το πώς ε, προχωρούν οι εργασίες. Είναι προφανές. οι εκπρόσωποι του ΕΛΚ θα πάνε. Θα πάνε και για προσωπικό... Υπό την προσωπική τους ιδιότητα βεβαίως, αλλά θα ενημερώσουν και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ο κύριος Φιέλνερ για την έκθεση. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι αυτή η έκθεση την οποία έλεγα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σας συστήνω να τη διαβάσετε. Εδώ και πέντε χρόνια είμαι στην ε, Επιτροπή αυτή και έχω διαβάσει πολλές ε, επικριτικές εκθέσεις από πλευράς ελεγκτικού συνεδρίου. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι αυτή είναι μία από τις πιο αυστηρές εκθέσεις που έχει έρθει ποτέ στα χέρια μας και περιέχει πάρα πολλές επικρίσεις. Θα, σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα. Γενικά όμως πρέπει να πω ότι η έκθεση για την δημόσια υγεία που έγινε η, μελέτη, ο έλεγχος που έγινε για αυτό το, τα προγράμματα δημόσιας υγείας είναι συγκεχημένα, δείχνουν τα πολλά προγράμματα ήταν συγκεχημένα, δεν ήταν ακριβή, έλειπαν λεπτομέρειες και στοιχεία απαραίτητα κλπ. κλπ. Εάν ε, είχα υποβάλει μια τέτοια έκθεση στο σχολείο μου, θα μου έλεγε ο δάσκαλος «Στόχευσες πολύ ψηλά και, όπως λέμε ελληνικά, έφευγε τα μούτρα σου». Ε, λοιπόν, εάν θέλουμε να μειώσουμε αυτές, ε, αυτό το πρόβλημα και δεδομένου ότι ο προπολογισμό δεν είναι τόσο πολύ μεγάλος για αυτά τα προγράμματα πρέπει να προσγειωθούμε και να μειώσουμε ε, αρκετά τις φιλοδοξίες μας. Είχε πάρα πολλούς φιλόδοξους και ευρύ στόχους αυτό το πρόγραμμα δημόσιας υγείας και έτσι γενικού στόχους χωρίς συγκεκριμένη εστίαση. Σε ορισμένου τομεί ε, δεν άρχισαν, δεν ξεκίνησαν προγράμματα καθόλου. Και ε, σε άλλες περιπτώσεις η Κομισιόν δεν μπόρεσε να, ε, να, να κάνει ένα σωστό έλεγχο και να δει αν ορισμένα προγράμματα που ξεκίνησαν επικαλυπτόντουσαν με άλλα προγράμματα που ήταν ήδη σε εξέλιξη. Γι' αυτό ακριβώς δεν δόθηκαν περισσότερες πιστώσεις στα προγράμματα δημόσιας υγείας, ενώ η Κομισιόν είχε ζητήσει ενίσχυση των πιστώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις προσπαθήσαμε να απειλήσουμε προβλήματα με ένα μικρό προϋπολογισμό. Σε άλλες περιπτώσεις όμως δεν μπορούμε να, να λύνουμε προβλήματα δίνοντας απλώς περισσότερα λεφτά. Υπήρχαν διαθρωτικά προγράμματα. Επίσης υπήρχαν στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί που δεν ήταν μετρήσιμοι. Δεν φτάνει χρόνος και δεν φτάνει το χρήμα για να λύσει τα προβλήματα προγραμμάτων που έχουν κολλήσει που δεν, δεν λειτουργούν. Πρέπει να έχουμε μετρήσιμα στοιχεία για να μπορούμε να κρίνουμε. Ποιο ήταν το όφελος των πιστώσεων που δόθηκαν, ποιο ήταν το όφελος των χρημάτων που επενδύσαμε και Βεβαίως, ορισμένοι τομεί δεν μπορούν να κρυθούν ε, με, ε, απλά ε, δεν είναι ασπρόμαυρα τα πράγματα ή άσπρα ή μαύρα. Υπάρχουν και γκρίζες περιοχές, γκρίζες ζώνες όπου χρειάζονται περισσότερα κριτήρια και περισσότερη έρευνα σε βάθος. Από ό,τι φαίνεται από την έκθεση αυτή, ε, το στοιχείο το οποίο ε, έχει το καλύτερο όφελος σε σχέση με το κόστος ήταν ε, ένα δίκτυο, ήταν το δίκτυο υγείας και αυτό το οποίο χρειάζεται στο μέλλον είναι πολύ καλύτερη παρακολούθηση και πολύ καλύτερη εστίαση, αλλά και ξεκάθαρους στόχους. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε το follow-up που χρειάζεται, ξεκάθαρους στόχους, οι οποίοι είναι και μετρήσιμοι, με μετρήσιμα κριτήρια μια μεγάλη, ένας μεγάλος κατάλογος που αναφέρει ε, στόχους και πολλαπλούς στόχους ε, δεν ωφέλει αν δεν μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε. Διότι ο τομέας δημόσιας υγείας είναι ευρύτατος και δεν πιστεύω ότι έχει νόημα στο μέλλον να, να, να ρίξουμε ακόμα περισσότερα λεπτά στις προβληματικές, ε, τα προβληματικά προγράμματα πριν έχουμε σαφή κριτήρια βάσει των οποίων μπορούμε να μετρήσουμε το αποτέλεσμα των επενδύσεων. Αυτά λοιπόν λέει η έκθεση επικριτικά. Πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα. Πρέπει η Κομισιόν να κάνει μία χαρτογράφηση, να καταγράψει ποια προγράμματα ε, ε, υπάρχουν, τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε, για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Επίσης, θα πρέπει να ερευνήσουμε λίγο περισσότερο Αξίζει τον κόπο να το κάνουμε αυτό. Ποια μέτρα αλλάζουν τη συμπεριφορά του κόσμου. Παραδείγματο χάρη, ε, μία έρευνα πιο επιστημονική για να δούμε ποια μέτρα μπορούμε να ενισχύσουμε που πραγματικά θα αλλάξουν την οτροπία και την, ε, ε, τη συμπεριφορά των πολιτών σε θέματα υγείας. Συγκεκριμένες δηλαδή δράσεις είναι ένα σοβαρό πρόβλημα η δημόσια υγεία και δεν μπορούμε να αφήσουμε το φάκελο, στο, να το κλείσουμε σε ένα σιρτάρι και να το αφήσουμε να σκονίζεται. Πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Ερικ Γκρετά, εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο εισηγητής σας συνόψισε καταπληκτικά την έκθεση του δικαστηρίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τι άλλο να πω. Είμαι απλώς στη διάθεση της Επιτροπής σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις για την έκθεση αυτή. Ουδής. Προχωρούμε. Έχουμε το επόμενο σημείο, το σημείο 15. Ειδική έκθεση 1-2009 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου τραπεζικά μέτρα στην περιοχή της Μεσογείου στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕΝΤΑ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ματιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόγραμμα ΜΕΝΤΑ ξεκίνησε το 1996 και τέλειωσε το 2006 ήταν το βασικό χρηματοδοτικό όργανο της Ένωσης για να υλοποιήσει την ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση. Το πρόγραμμα τελείωσε το 2006 και πέρασαμε στο νέο εργαλείο που ήταν ε, το εργαλείο ε, γειτονίας. Ε, μέχρι το 2000 με το 2006 ε, είχαμε 536 ε, εκατομμύρια, ενώ προηγουμένως 424 εκατομμύρια. Επίσης προσπαθήσαμε να δούμε αν υπήρξε παρακολούθηση από την ε, Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είχαμε τρεις τραπεζικές δραστηριότητε. Τεχνική αρρωγή και επιδότηση, επιδοτούμενα επιτόκια και επιχειρήσεις κεφαλαίων κινδύνου. Για 30 προγράμματα, 24 υλοποίησαν τους στόχους, ενώ τα 6 υλοποιήθηκαν μερικά. Σαν παραδείγματα επιτυχημένα ήταν τα... η μικροχρηματοδότηση και η ανάπτυξη στην Τινησία και στο Μαρόκο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τα επιδοτούμενα ε, επιτόκια και τα κεφάλαια κινδύνου, τα αποτελέσματα είναι πιο μετριασμένα, αρκετά ικανοποιητικά. Ε, υπάρχουν ελλείψεις στις πληροφορίες και καθυστερήσει ορισμένα προγράμματα. Ένα πρόγραμμα που είχε σαν σκοπό να μειώσει τη μόλυνση στο κόλπο της, του Γκαμπέ στην Τινησία το 1999 είχε εγκριθεί, αλλά δεν ξεκίνησε παρά μόνο πολύ αργότερα. και οι εργασίες που θα είχαν αρχίσει το 2002 ε, αναβλήθηκαν για το 2009 και 2010. Θα ήθελα να επίσης την προσοχή της Επιτροπής στο να, στην ανάγκη να υπάρχει αποτελεσματικό συντονισμός μεταξύ της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Κομισιόν και άλλων διεθνών εταίρων. Θα πρέπει να ανταλλάσσονται πληροφορίες τακτικά σε τοπικό επίπεδο, ούτως ώστε να υπάρχει συμπληρωματικότητα και συνοχή. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, διαπιστώνουμε ότι η εποπτεία δεν ήταν επαρκή στα πρώτα χρόνια του προγράμματος, ιδίω στις περιπτώσεις όπου η Κομισιόν βασιζόταν αποκλειστικά στην παρακολούθηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πριν το 2005, θα ήθελα ε, να προχωρήσουμε γρήγορα ε, για να υπογραφούν τα τελευταία έγγραφα μεταξύ της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Για την παρακολούθηση των τραπεζικών επίσης δραστηριοτήτων θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε αυτό το επίπεδο, τώρα στα πλαίσια του νέου εργαλείου ε, γειτονίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ίγκορ Λούμπντορς, εκπρόσωπος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, Uh, Νομίζω ότι η συγγήτριά σα, η κυρία Ματιέ, έκανε μια έξωση, έξοχη σύνοψη, την οποία παρουσιάζει και στα έγγραφα εργασίας που σας έχει δώσει. Αν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις θα μπορούσα να σας απαντήσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Sí, gracias, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ την κυρία Ματιέ για την έκθεση που μας παρουσίασε. Έχω κάποιες ερωτήσεις, κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το πώς λαμβάνοντας υπόψη και τα διάφορα μέτρα στα οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα ΜΕΝΤΑ και τους ε, διάφορες δείκτες αποτελεσματικότητας, ε, πώς ε, λάβαμε τις αποδείξεις. Μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και υπήρχαν κάποιες αδυναμίες περιβαλλοντικά θέματα εντοπίσαμε θετικά και αρνητικά στοιχεία και δεν υπάρχουν κοινωνικά στοιχεία στους δείκτες που μετρήσαμε. Σε άλλα ταμεία, όπως ακούσαμε χθες, μετράμε την αποτελεσματικότητα και σε σχέση με την ε, ε, μετατροπή του κοινοτικού ιστού, του οικονομικού ισιού, κυρίως όσον αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν, ε, αν μπορεί να μου πει η κυρία Ματιέ, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη, προκειμένου να δώσουμε συστάσεις ε, ε, για αυτό το μέσο εταιρικής σχέσης και γειτονίας και θα ήθελα να ρωτήσω και το ελεγκτικό συνέδριο με ποιο τρόπο αυτές όλες οι πτυχές ε, που είχαν ε, καθοριστεί ότι θα μελετηθούν στην εντολή ε, θα ληφθούν υπόψη. Τα αποτελέσματα που λάβαμε, πώς τα ρυθμίζουμε σε θέματα παρατυπιών, μας ενδιαφέρουν και τα καλά αποτελέσματα, ε, οι αλλαγές που έγιναν σε χώρες οι οποίες εφαρμόστηκαν κοινωνική υφή, ε, αναγνώριση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ευχαριστώ. Κυρία Ματιό θα απαντήσει. Όταν ε, επισκεφθήκατε αυτές τις χώρες ε, στις αποστολές σας, θα έχετε διαπιστώσει, το είπα βέβαια κιόλα, ότι τα προγράμματα δεν είναι επικεντρωμένα. Είναι πάρα πολύ διασπαρμένα. Τα προγράμματα, για να το πω έτσι, είναι κατακαιρματισμένα. Δεν υπάρχει πραγματική πολιτική που να περνάει μέσα από τα προγράμματα. Θα μπορούσαμε όντως να συστήσουμε στην Κομισιόν να προωθήσει μια πραγματική πολιτική και περιβαλλοντική βέβαια. Αλλά ούτως ή άλλως τα περιβαλλοντικά προγράμματα συμπεριλαμβάνουμε και μια κοινωνική διάσταση. Επομένως, αυτό που είπατε είναι απόλυτα σωστό. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Το χρειαζόμαστε άλλωστε όταν συζητάμε σχέσεις με τη Μεσόγειο. Αλλά στην προηγούμενη θητεία κάποια στιγμή αυτό προέκυψε από κάποιες ε, αποστολές και κάποιες αντιπροσωπείες ε, οι οποίες μετέβησαν εκεί ε, από πλευράς Επιτροπή μας. Προέκυψε η ιδέα να υπάρχουν στις κοινοβουλευτικές αποστολές, όταν γίνονται τέτοιες αποστολές, να υπάρχει ένα μικρό ερωτηματολόγιο, όχι υποχρεωτικό γιατί δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανένα, ώστε οι αντιπροσωπείες που επισκέπτονται κάποια χώρα, δεδομένου ότι πάνε και με δαπάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσθέσουν και κάποιες ερωτήσεις, δηλαδή αν μπορούσαμε να τις παρακαλέσουμε να προσθέσουν ε, κάποιες ερωτήσεις για να τις έχουμε ως στοιχείο μελέτης, διότι δεν μπορούμε να επισκεφθούμε όλες τις χώρες, αλλά να δούμε τι γίνεται με αυτές τις νέες μορφές βοήθειας, κυρίως αυτό το μέσο γειτονίας. Δεν ξέρω αν ο πρόεδρος θεωρεί ότι είναι υπερβολικό, αλλά οι ίδιες οι αντιπροσωπείες μας είχαν πει στο παρελθόν ότι όταν επισκέπτονταν ε, κάποια ε, μέρη στα οποία υπήρχαν προγράμματα τα οποία είχαν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν ίσως να δώσουν κάποια στοιχεία και εδώ στην Επιτροπή μας είναι ο χώρος για να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Ο κύριος Σοντή. Ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ματιέ για την παρουσίαση που μας έκανε και να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο που ενδιαφέρεται για τις τραπεζικές δραστηριότητες. Ευχαριστώ και το ελεγκτικό συνέδριο γιατί είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο θέμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εδώ και χρόνια ζητάμε αυτό το χρηματοδοτικό μέσο να αποτελέσει τμήμα οικονομικής ρύθμισης, χρηματοδοτικής ρύθμισης. Το ζητάμε χρόνια και το ζητάμε και φέτος. Θα δούμε τι θα γίνει. Είχα ζητήσει στο παρελθόν το ελεκτικό συνέδριο να εξασφαλίσει ένα ρόλο επαγρύπνησης ό,τι αφορά τους οικονομικούς κανόνες. Και μου είπαν ότι το ε, ελεκτικό συνέδριο δεν κάνει τέτοιου είδους εποπτεία για τα τραπεζικά θέματα. Ε, για τις ε, επιχειρήσεις που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως θα μπορούσε το ελεκτικό συνέδριο να παίξει κάποιο ρόλο. Βέβαια είναι πολύ περίπλοκα θέματα. Ίσως λοιπόν ε, θα μπορούσα να κάνω μια πρόταση. Είχαμε προτείνει να υπάρξει μια ευρωμεσογειακή τράπεζα στην... Ε, θα μπορούσαμε να ακούσουμε αν έχει νόημα να έχουμε μια πραγματική, τράπε... να έχουμε μια πραγματική τράπεζα. Παρά να περνάμε μέσα από όλα αυτά τα μέσα, το, το ΜΕΝΤΑ ε, ή το ΦΕΜΙΠ, αυτό το Ταμείο Υποστήριξης, το ΦΕΜΙΠ, Περνάμε δηλαδή μέσα από όλα αυτά τα πράγματα, αντί να έχουμε μια πραγματική τράπεζα. Έχει νόημα να έχουμε λοιπόν μια πραγματική τράπεζα. Θα επανέλθω τώρα σε αυτή την ιδέα της, ε, των κανόνων, των ε, οικονομικών κανόνων για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Κεντρική Τράπεζα διστάζει, δεν υπάρχει πολιτική βούληση στο εσωτερικό του Συμβουλίου. Βλέπουμε, με βάση τις πληροφορίες που μας λέει το ελεγκτικό συνέδριο για αυτό το μικρό τμήμα δραστηριοτήτων ευρωμεσογειακού χαρακτήρα. Βλέπουμε λοιπόν πόσο χρήσιμο είναι να συνεχίσουμε να απαιτούμε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να έχει χρηματοδοτικούς κανόνες, οικονομικούς κανόνες, γιατί είδαμε μια κάποια ταξία. Τα πράγματα μπαίνουν σε κάποια τάξη, αλλά παρόλα αυτά χρειαζόμαστε μια ρύθμιση θα πρέπει να ελέγχουμε τις οικονομικές ε, δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που είναι δική μας αρμοδιότητα της ε, Επιτροπής μας. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να επαγρυπνούμε για τις ε, οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτό δεν είναι εύκολο γιατί είναι διακυβερνητικό εργαλείο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. και δεν έχουμε τελικά νομική αρμοδιότητα. Αλλά ο πρόεδρος, ο οποίος είναι θαυμάσιος άνθρωπος, είπε ότι θα προσέχει ιδιαίτερο τις θέσεις των βουλευτών. Το πρώτο μας καθήκον ποιο είναι, να ελέγχουμε τα μέσα, τα εργαλεία. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγορώ. Αλλά τη στιγμή που η Επιτροπή αποφασίστηκε να βασιστεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για διάφορα μέσα και εργαλεία τα οποία συγχρηματοδοτούμε, είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε οικονομικά την, ε, τις δραστηριότητες της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είμαι απόλυτα πεπισμένος λοιπόν ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα. Συμφωνώ απόλυτα. Ούτω ή άλλω αυτό είναι στα καθήκοντα τη Επιτροπή μα ε, να ελέγχουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 16. Eh, Έχουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ο οποίος θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ. Δύο λόγια θέλω να, μιλ... να πω και εγώ εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέγομαι Έχω άλλο όνομα, δεν είμαι αυτός ο κύριος που είπατε, ο κύριος Ντεκαμπαγιέρα. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Ματιό για την έκθεσή της, καθώς και το ελεγκτικό συνέδριο. Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του ελληνικού συνεδρίου και της κυρίας Ματιό. Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η περίοδος που ελήφθη υπόψη από το ελεγκτικό συνέδριο και αυτό είναι φυσικό, μια και είναι υποχρεωμένο να ελέγξει αυτό που τελείωσε για να κρίνει τις επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν το διάστημα ε, είναι πολύ προγενέστερο από την σημερινή περίοδο. Και επειδή τα πράγματα κινούνται πολύ, είναι σαφές ότι η σημερινή κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με την περίοδο για την οποία μιλάμε. Επομένω, το επίπεδο Εποχοπτίας και επαγρύπνησης των επιχειρήσεων σήμερα είναι πολύ πιο υψηλό από ό,τι ήταν στο παρελθόν, από ό,τι ήταν σε αυτή την περίοδο. Έχουμε και μια ειδική μονάδα εξειδικευμένη που παρακολουθεί αυτές τις ε, επιχειρήσεις ε, διευκόλυνση των επενδύσεων. Το FEMIP δεν, υπάρχει, δεν είναι το μοναδικό εργαλείο. Δημιουργήθηκαν και άλλα εργαλεία και άλλα μέσα. Έχουμε λοιπόν ειδικού που παρακολουθούν τα πράγματα καθημερινά και με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο και αυστηρό τρόπο. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η ίδια δημιούργησε επιτόπια γραφεία σε πολλές ε, μεσογειακές χώρες, επομένως σε επίπεδο τοπικού συντονισμού, παρακολούθησης ε, των επιχειρήσεων, ε, λιεζών, σχέση με τα γραφεία μας. Είμαστε πολύ πιο κοντά, έχουμε μια συνεργασία δηλαδή και ένα συντονισμό και έναν αποτελεσματικό έλεγχο πολύ πιο αυστηρό και σας καθησυχάζω ότι υπάρχει ένας, μια πανοπλία δικτών επιδοτήσεων, επιδόσεων συγγνώμη, που υλοποιούμε και εμείς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι εκθέσεις αξιολόγησης. Γιατί πολύ σωστά είπε η κυρία Αγέλα και ο κύριος Σοντή, αν αυτές οι προσπάθειες δίνουν αποτελέσματα, λοιπόν, σας ε, καθησυχάζω ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης ε, τις οποίες θα σας στείλουμε, για όλα τα εργαλεία του ΜΕΝΤΑ 2, θεωρούν ότι όλες οι επιχειρήσεις που υλοποιήθηκαν είναι θετικές και στα κεφάλαια κινδύνου και στα επίπεδο της ε, ε, επιδότησης των επιτοκίων. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι μελέτες γίνονται από εξωτερικά γραφεία χωρίς παρέμβαση της Κομισιόν. Επομένως, την έκθεση θα την δείτε και νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία που θα διαβάσετε θα σας καθησυχάσουν. Τώρα, για την κοινωνική διάσταση. Υπενθυμίζω ότι τα περιβαλλοντικά προγράμματα και τα προγράμματα επικίνδυνου κεφαλαίου έχουν και μια κοινωνική διάσταση γιατί δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης. Τα προγράμματα δεν είναι μόνο οικονομικά. Αν αντιμετωπίζουμε όλα τα κοινωνικά προβλήματα, αν δίνουμε πόσιμο νερό ε, ή καλύτερο νερό, καλύτερης ποιότητα σε μια περιοχή, ε, προφανώς ε, βελτιώνουμε το περιβάλλον, αλλά και την ποιότητα ζωής του πληθυσμού. Επομένως, νομίζω ότι είναι πολύ αφαιρετικό να θεωρήσουμε ότι τα προγράμματα ε, απλώς ε, προωθούν τον τίτλο τους. Ναι, προφανώς είναι κεφάλαια κινδύνου, αλλά υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα λοιπά. Ναι, περιβαλλοντικά προγράμματα, αλλά πίσω από αυτά υπάρχουν πληθυσμοί που έχουν ανάγκη από πόσιμο νερό, καλό νερό, ε, επεξεργασία των λιμάτων κτλ. Για την παρατήρηση του κυρίου Οντί, για τις οικονομικές ρυθμίσεις, τους οικονομικούς κανόνες. Οι επιχειρήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Επενδύσεων ε, είναι επιχειρήσεις στις οποίες συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Θα ήθελα να κάνω ένα προσωπικό τώρα σχόλιο. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα ανά τον κόσμο τέτοιου τύπου και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λειτουργεί πάρα πολύ καλά, συνεργαζόμαστε καλά μαζί μας, είναι πολύ σοβαρό σοβαρός φορέας. Επίσης δουλεύουμε με τους ε, χρηματοδοτικούς φορείς των κρατών μελών, η ΑΕΦΔ, η γερμανική, η ισπανική, ισπανικές ε, υπηρεσίες και πριν ε, δημιουργήσουμε νέους φορείς πρέπει να σκεφτούμε ότι για τις διαπραγματεύσεις χρειαζόμαστε μήνες αν όχι χρόνια. Και συχνά το πρώτο αποτέλεσμα είναι ότι σταματάμε να δουλεύουμε σε μια πρώτη φάση. Καλό είναι να είμαστε πιο ταπεινοί, πιο συνετοί και απλώς να βελτιώσουμε αυτά που έχουμε ήδη και αυτό που κάνουμε ήδη. Να βελτιώσουμε το σύνολο των μέσων και εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Νομίζω είναι πιο σωστό. Σας ευχαριστώ. Ο... Το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κανονικά, δεν θα ξαναζητούσα το λόγο για την ίδια έκθεση, αλλά πιστεύω ότι ένα στοιχείο πρέπει να, να διευκρινιστεί. Το ελεγκτικό συνέδριο διαλέγει τα καλύτερα δείγματα, έτσι ώστε να μπορούμε να κρίνουμε τι έχει γίνει. Θέλω λοιπόν να κάνω μία να ξεχωρίσω αυτά τα οποία έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν και τη σημερινή κατάσταση. Η πρακτική του ελεγκτικού συνεδρίου είναι μετά από δύο χρόνια να επανέρχεται σε ένα φάκελο, να ξανανοίγει ένα φάκελο και να κάνει μία ανασκόπηση του τι έχει γίνει από τότε που έγινε ο έλεγχος και να ενημερώνει το φάκελο για την ε, τρέχουσα κατάσταση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Κύριε Γελασέντε. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να επανέλθω για άλλη μια στιγμή σε αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, τον οποίο ευχαριστώ για τα σχόλια και τις πληροφορίες. Αλλά κάτι δεν κατάλαβα. Καταλαβαίνω βέβαια πάρα πολύ καλά και είναι σαφές ότι μια διαδικασία εξυγίανσης των υδάτων κλπ. έχει και κάποιε κοινωνικέ επιπτώσει, αλλά κάπου είτε το ελεγκτικό συνέδριο είτε οι πληροφορίες που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εντολή ήταν να δούμε αν υπάρχουν ε, ε, παρατυπίες ή αν όλα εντάξει ή αν υπάρχει καλή εφαρμογή από πλευρά ε, χρηματοοικονομικής, κυρίως εφαρμογή των κονδυλίων των ταμείων, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μελετήσουμε και τα αποτελέσματα. Δηλαδή, είναι ισορροπημένα τα δύο πράγματα. Ε, ναι, μεν μας λέτε ότι προφανώς υπάρχουν και κοινωνικές επιπτώσεις, αλλά κάπου δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ή δεν σταθήκαμε σε αυτές. Διότι αυτό που μας ενδιαφέρει και εμένα με ενδιαφέρει ως Κοινοβούλιο, όταν κάνουμε μια ανακοίνωση προς τα έξω, να μην λέμε απλά ότι όλα τα τιμολόγια ήταν εντάξει, πήραμε όλα τα λεφτά μας και ε, ε, που δεν είχε, αυτά που δεν είχαν δαπανεθεί τα πήραμε πίσω αλλά και ότι υπήρχαν κάποιε συνέπειε, δημιουργήθηκαν θέσεις απασχόλειας. Κάπου πρέπει να εμφαίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν θα είναι στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου ή στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας λέτε ότι στο ΜΕΝΤΑ 2 θα μα προσφέρετε αυτή την αξιολόγηση, αλλά μα ενδιαφέρει ω κοκομπού να έχουμε και αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, έγινε μια καλή οικονομική εφαρμογή αξιολόγηση ε, του έργου κλπ, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να ξέρουμε και ότι οι στόχοι της συνεργασίας, της ανάπτυξης, κυρίως ε, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, καλύπτονται. Θέλουμε δηλαδή κάπου να μας δίνονται και αυτές οι πληροφορίες για να έχουμε όλα τα στοιχεία και να μπορούμε να τα διαβάσουμε κιόλας. Grazie. Ευχαριστώ. Ωραία. Να περάσουμε στο σημείο 15 ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, αριθμός 5 του 2009, διαχείριση των ταμιακών διαθεσίμων τη επιτροπή Ο κύριο Ήταλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό, αυτή είναι μια έκθεση που αφορά την οικονομική διαχείριση της Κομισιόν. Έγινε ο έλεγχος για να δούμε εάν η Κομισιόν συμμορφώνεται με τους κανόνες της οικονομικής διαχείρισης και αν έχει συστήσει δικούς της εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου. Όσον αφορά λοιπόν την οικονομική διαχείριση, εμπλέκονται δύο γενικές διευθύνσεις, ε, Γενική Διεύθυνση Budget και Προϋπολογισμού και Γενική Διεύθυνση Exin. οι ελεγκτές οι οποίοι συνέταξαν αυτή την θαυμάσια έκθεση και του συγχαίρω σημείωσαν τα εξής. Γενικά η Εκτελεστική Επιτροπή έχει εφαρμόσει τα πιο σημαντικά στοιχεία της νομοθεσίας Υπάρχουν όμως ορισμένες παρατηρήσεις. Καταρχάς, η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού, αντίθετα από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ, δεν έχει συντάξει μία έκθεση που να αναφέρει τα συστήματα διαχείρισης ρίσκου, risk management. Πρέπει λοιπόν να υποβάλει καλύτερη τεκμηρίωση για το πώς διαχειρίζεται τα ρίσκα, τους κινδύνους. Και το πιο σημαντικό σημείο είναι, πιο σημαντική παρατήρηση είναι ότι αυτές οι δύο γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν δεν έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους για την εφαρμογή και εποπτεία μιας κοινή στρατηγικής διαχείρισης ρίσκου. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μία από τις δύο διευθύνσεις αποφάσισε να έχει ένα απόθεμα ε, σε μια τράπεζα για τη διαχείριση κινδύνου, το οποίο δεν ακολούθησε η άλλη διεύθυνση. Δεν έχει λοιπόν υπάρξει συντονισμός μεταξύ των δύο διευθύνσεων και λέει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ότι το οικονομικό ρίσκο θα πρέπει να μελετάται και να υποπτεύεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και θα πρέπει η διαχείριση του κινδύνου να βασίζεται σε μία συγκερασμένη πολιτική διαχείρισης έτσι ώστε κάθε φορά και αν εντοπίζονται προβλήματα να μπορεί αμέσως να υποβληθεί μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συστήνει το ελεγκτικό συνέδριο να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο γενικών διευθύνσεων ώστε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση και εποπτεία της διαχείρισης του ρίσκου, των κινδύνων δηλαδή. Μία άλλη παρατήρηση αφορά τις ποινές, τις ε, ποινές ε, που εφαρμόζονται, που ισχύουν στους τραπεζικούς ε, λογαριασμούς και προτείνει να αλλάξει η κατάσταση και η Γενική Διεύθυνση Budget έχει υιοθετήσει μια νέα απόφαση για να βελτιώσει την ασφάλεια των τραπεζικών λογαριασμών της. Ευχαριστώ κύριε Ήταλα. Να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου, τον κύριο Λούβροτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη, πιστεύω μετά από αυτά που άκουσα από τον κύριο Ήταλα, ότι συνόψισε με σαυμάσιο τρόπο την έκθεση αυτή για την διαχείριση των οικονομικών της Κομισιόν. και είμαι στη διάθεσή σας ε, για να απαντήσω σε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις που τυχόν έχετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίασή του και το ελεγκτικό συνέδριο για αυτή την έξοχη έκθεση. Θα ήθελα να θέσω και μία ερώτηση. Στα πλαίσια της Κοκομπού διαπιστώσαμε τους ε, ταμιακούς λογαριασμούς ε, οι οποίοι ρυθμίστηκαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκαναν κάποιες ε, προτάσεις, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή τη δυστυχή περίσταση, στους ελέγχους σας. Ε, διαπιστώσατε ότι υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί εκτός προϋπολογισμού ή όλα τα ταμιακά διαθέσιμα είναι εντός προϋπολογισμού. Αυτή είναι η ερώτησή μου η πρώτη. Η δεύτερη ερώτηση στα πλαίσια των ρυθμίσεων η λειτουργία των ταμιακών δαθεσίμων γίνεται βάση ε, λογιστικών ελέγχων. Οι διεθνείς ε, λογιστικοί κανόνες προβλέπουν ο λογιστής να μην κρατάει τους λογαριασμούς των ταμιακών διαθεσίμων. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι ε, ε, άποψη έχετε για την ε, οργάνωση αυτή που προβλέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό, διότι ο δημοσιονομικός κανονισμός δίνει αυτή την εξουσία στο λογιστή. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι άποψη το ελεγκτικό συνέδριο. Ο λογιστής ο οποίος είναι υπεύθυνο για τα ταμιακά διαθέσιμα θα πρέπει να ασχολείται και με αυτούς τους λογαριασμούς. Παρακαλώ, εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τους ελέγχους προϋπολογισμού, όλων των προϋπολογισμών, δεν ήταν στόχος μας να ελέγξουμε ε, όλους τους λογαριασμούς και την ε, διαχείρισή τους, εμείς θέλουμε να ελέγξουμε το σύστημα ελέγχου της Κομισιόν. Γενικά το σύστημα ελέγχου όλων των οικονομικών και όλων των λογαριασμών της Κομισιόν είναι ικανοποιητικό. Υπάρχουν ορισμένες πτυχές που μπορούν να γίνουν καλύτερες, να βελτιωθούν. Όσον αφορά τώρα τα λογιστικά ε, στοιχεία και την ε, διάθεση την ενημέρωση των ταμιακών διαθεσίμων, πιστεύω ότι τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζει ο έλεγχος μας συμφωνούν με αυτά τα οποία εφαρμόζει η Κομισιόν. Δηλαδή, η Κομισιόν εφαρμόζει σωστά τα κριτήρια λογιστικού ελέγχου. Και οτιδήποτε μικρές ε, παρατυπίες έγιναν ε, θα διορθωθούν ε, σύντομα. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Prego. Diamo la parola al rappresentante della Commissione. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Mm. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως για να απαντήσω στον κύριο Ντί Η κατάσταση στην οποία αναφέρθηκε έχει ρυθμιστεί εδώ και κάποιους μήνες ε, και να σας ε, καθησυχάσω και για το διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των ε, λογιστών και των ταμιακών διαθεσίμων. Αυτός ο οποίος διαχειρίζεται τους λογαριασμούς και αυτός που τους ελέγχει είναι προφανώς διαφορετικά πρόσωπα. Τώρα, Έγιναν κάποιες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των υπηρεσιών του ελεκτικού συνεδρίου. Οι συστάσεις ε, οι οποίες ε, αναφέρεται ακολουθούνται πάρα πολύ επισταμένα ε, και κυρίως έχουμε σταθεί σε θέματα ανάλυσης κινδύνου και της ανακοίνωσης της ανάλυσης κινδύνου στην Κοκομπού. Αυτά άλλωστε έχουν γίνει, διότι βρίσκονται και στο σημείωμα το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή σας, διαβιβάζεται κάθε 1η Απριλίου και επίσης και στην ετήσια έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης ε, Προϋπολογισμού, η οποία είναι διαθέσιμη στη γραμματεία της Κοκομπού και τη δίνουμε στις αρχές του χρόνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ταβέχ. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στην επόμενη έκθεση. Έκθεση αποδοτικότητα της δαπάνης των διαθερωτικά μέτρων για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων κατά της περίοδου προγραμματισμού 1994-1999 και 2000-2006. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ντόιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Όπως ε, ήδη έχει δηλώσει ο πρόεδρος, αυτό το έγγραφο εργασίας αφορά τη διαχείριση των πιστώσεων για τα προγράμματα τα διορθωτικά σε αυτές τις δύο χρονικές περιόδους. Καταρχάς, του χρόνου, στο Sheffield, στο Ενωμένο Βασίλειο, ξεκίνησε η λειτουργία της πρώτης, ομάδας, της πρώτης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων. Είναι η 50η επέτειος, 50 χρόνια, πριν από 50 χρόνια λειτουργήσε αυτή ομάδα. Ε, συγγνώμη, μονάδα. Και επειδή στην ε, Μεγάλη Βρετανία είχε σημειωθεί μια μεγάλη οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη, υπήρχε αυτή η ανάγκη σωστή διαχείρισης των αποβλήτων. Κυρίες και κύριοι, το ελεγκτικό συνέδριο μας παρουσίασε μια αξιόλογη έκθεση και ε, από πλευράς μου ευχαριστώ ε, το ελεγκτικό συνέδριο και τους δύο συναδέλφους που συνέταξαν την έκθεση αυτή είναι εξαίσθηση υψηλής ποιότητας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ταμείο Συνοχής και από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης γίνεται συγχρηματοδότηση για τις ε, μονάδες διαχείρισης αποβλήτων. Στο πρόγραμμα 2000-2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνησε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Έδωσε δηλαδή ως ενίσχυση και μετα τώρα στο καινούριο πρόγραμμα 2007-2013 αυτό το στοιχείο είναι 13 εκατομμύρια ευρώ μόνο. είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα αυτά. Είναι λιγότερο από το μισθό, τον ετήσιο μισθό ενός ενός ποδοσφαιριστή. Ψυχία δηλαδή. Σε όλη αυτή την περίοδο μέχρι το 2006, όπως σας είπα, ξοδεύτηκαν πάνω από 10 δις, 10 δις, όχι εκατομμύρια, 10 δις, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα και γι' αυτό η ειδική έκθεση αυτή του ελεγκτικού συνεδρίου ε, ασχολείται και αναφέρει συγκεκριμένα τα προγράμματα αυτά στις τέσσερις χώρες. Έκανε ελέγχους στις μονάδες αυτές, έλεγξε τους φακέλους, ε, την τεκμηρίωση ε, στις μονάδες και κάνει τρεις συστάσεις βάσει των συμπερασμάτων. Πρώτον, δεχόμαστε και σημειώνουμε αυτά τα οποία λέει το ελεγκτικό συνέδριο. Πρέπει να πιέσουμε και να κινητοποιήσουμε τις αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν το 100% δυναμικό αυτών των μονάδων διαχείρισης αποβλήτων που έχουν συγχρηματοδοτηθεί. Να χρησιμοποιούν δηλαδή το πλήρες δυναμικό όπως λέει το ελεγκτικό συνέδριο, σε ορισμένε περιπτώσεις οι μονάδες αυτές που έχουν κατασκευαστεί δεν χρησιμοποιούνται στο 100%. Υπάρχει λοιπόν περισσότερη δυνατότητα διαχείρισης αποβλήτων, μεγαλύτερου όγκου. Επίσης, ορισμένες μονάδες προσβλέπουν σε μελλοντικές επενδύσεις για να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις. Όταν όμως μια εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων δεν χρησιμοποιείται στο 100% πριν κάνει οποιαδήποτε επέκταση, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσει το 100% των δυνατοτήτων της. Και η, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία καλύπτει την διαχείριση της ηλίως, της λάσπης των λιμάτων χρονολογείται από το 1986 και η Κομισιόν έχει δηλώσει ότι ήδη εργάζεται στην, για την ανασεώρηση αυτής της οδηγίας Διαχείριση της λάσπης ε, έχει περάσει, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια ή πολλά λίματα και πρέπει εν πάση περιπτώσει να αναθεωρηθεί αυτή η οδηγία. Διότι η χρήση της λάσπης, της ηλίως αυτής των λιμάτων είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, προσφέρει πολλές δυνατότητες και θα πρέπει να επικαιροποιηθεί αυτή η οδηγία. Σε αυτό το έγγραφο εργασίας έχω κάνει και εγώ μια πρόταση. Οι εγκαταστάσεις ε, διαχείρισης ε, λιμάτων που ήδη λειτουργούν πρέπει να λειτουργούν απολύτως αποδοτικά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν, όταν γίνεται ένας μειοδοτικός ή προκυρήσει ένα διαγωνισμό για έργα, για εγκαταστάσεις, θα πρέπει να συντάσει, ε, να έχει διάφορα κριτήρια ελέγχου αλλά και κατευθυντήριες γραμμές συγκεκριμένες, ώστε η αξιολόγηση λειτουργίας ε, των εγκαταστάσεων αυτών να είναι απολύτως ε, ικανοποιητική, να γίνεται δηλαδή με τον καλύτερο τρόπο. Το ελεγκτικό συνέδριο διαπίστωσε επίσης ότι τα έργα αυτά θα πρέπει να κρίνονται πιο με πιο αυστηρά κριτήρια, έτσι ώστε οι τελειωμένες εγκαταστάσεις να μην έχουν αυτό το έλλειμμα δυναμικού, δηλαδή να λειτουργούν στο 100%. Αυτά, Πρόεδρε, είχα να πω συνοπτικά ε, για την παρουσίαση της έκθεσης αυτής. Τώρα ο εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου, Ουβίδιου Ισπύρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, της Επιτροπής Ελέγχου το έγγραφο εργασίας το οποίο παρουσίασε ο κύριος Ντόιτς, ο οποίος είναι και ειδικό εισηγητής επί της εκθέσεως του ελεγκτικού συνεδρίου, συνόψισε πάρα πολύ καλά την έκθεσή μας. Αυτό το οποίο θέλω να επαναλάβω χωρίς να ε, ε, αυτό που θέλω να προσθέσω, χωρίς να επαναλάβω αυτά που είπε, είναι το εξή. Η δημοσίευση αυτής της ε, εκθέσεως έγινε δεκτή με μεγάλη ικανοποίηση. Είχε μάλιστα θετικό αντίκτυπο στον τύπο, ε, στα μέσα ενημέρωση και τον ενέκριναν και, και πολύ ακαδημαϊκοί δεδομένο ότι άπτεται και τον ελέγχων σε θέματα περιβάλλοντος. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας αυτός η διαχείριση των ε, λιμάτων για τους Ευρωπαίους πολίτες και πιστεύω ότι η έξεση αυτή με τα συμπεράσματα όπως θα υιοθετηθεί από εσά θα συμβάλλει περαιτέρω στις προσπάθειές μας βελτίωσης προστασίας του περιβάλλοντος και θα ενεργήσει προς το συμφέρον των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον κύριο Ντόιτς για την εξαιρετική έκθεσή του. Ήθελα απλώς να ρωτήσω, προκειμένου να εμβαθύνουμε και λίγο, γιατί θεωρώ ότι τα θέματα είναι σημαντικά, σημεία που αφορούν τις αδυναμίες του εφαρμοστέου συστήματος. Μπορεί να είναι και το πιο εξαιρετικό ή το πιο ευνοϊκό, αλλά πάντα φαίνεται το πρόβλημα της έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης, ε, της έλλειψης εμπειρογνωμόνων ή και τεχνικής εμπειρίας των, τεχνικών, ε, των ε, τοπικών αρχών. Συγγνώμη. Η εφαρμογή μιας οδηγίας υποχρεώνει σχεδόν όλους τους Δήμους να θέσουν σε εφαρμογή έργα για τον καθαρισμό των λιμάτων. Πολλές φορές τα έργα αυτά είναι πολύ μεγάλα, ε, υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει σύνδεση με το σύνηθε σύστημα αποχέτευσης ή τον, το σύστημα από τον οποίο φτάνουν τα ύδατα. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα λοιπόν με τη διασύνδεση εκεί και θα ήθελα το ελεγκτικό συνέδριο να μας διευκρινίσει λίγο καλύτερα το θέμα αυτό και το κατά πόσο θα μπορούσαμε να προτείνουμε και μια μελέτη ε, για την έλλειψη εμπειρογνωμοσύνη, την έλλειψη τεχνικής γνώσης ε, των ε, τοπικών αρχών ε, για θέματα που αφορούν εφαρμογή ευρωπαϊκών κονδυλίων και είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το περιβάλλον. Θα ήθελα επίσης να μου διευκρινίσει το ελεγκτικό συνέδριο το θέμα των τιμολογίων. Υπάρχει κάποια σύσταση, υπάρχει κάποια ενημέρωση για το πώς προχωράει η εφαρμογή των ταμείων, αν έχουν ξεκινήσει τα εργοτάξια, τα σχέδια, αν υπάρχει αρκετή σοβαρότητα, αν είναι θετικά τα στοιχεία, αλλά υπάρχει επίσης και το θέμα της διασφάλισης της ε, συντήρησης αυτών των έργων. Δεν μιλάμε μόνο για ε, προγράμματα καθαρισμού λιμάτων, για παράδειγμα, μιλάμε για γενικότερα συστήματα. Πέραν από τις συστάσεις λοιπόν που μας δίνονται εδώ, θα μπορούσατε να εμβαθύνετε λίγο περαιτέρω στο θέμα. Με ποιον τρόπο μπορούμε να δούμε τις ανάγκες που υπάρχουν στα μελλοντικά προγράμματα και αν θέλετε θα μπορούσατε να μας απαντήσετε και τι γίνεται με αυτά τα σχέδια τα οποία θέλουν και μια κάποια ε, εφαρμογή, ξεκινούν πάρα πολύ καλά αλλά υπάρχει αυτή η έλλειψη και κάποια στιγμή μπορεί να σταματήσει η λειτουργία τους ή να υπολειτουργούν για δύο λόγους ή γιατί δεν υπάρχουν αρκετές ε, δυνατότητες τεχνικές των ε, ε, τοπικών αρχών ή γιατί δεν υπάρχουν ε, αρκετά κονδύλια για τη διατήρηση των, ε, των δικτύων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Στην Ιταλία, μεταξύ των βασικών προβλημάτων με τη διαχείριση των κοινοτικών κονδύλιων είναι ακριβώς το θέμα του καθαρισμού των υδάτων. Αυτό έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δημιουργεί μόλυνση επίσης ε, και έχουμε ε, πρόβλημα με κακή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Με αυτόν τον τρόπο διασπαθίζονται εκατοντάδες ε, χιλιάδες ευρώ. Εξάλλου η Όλαφ ενημερώθηκε γι' αυτό. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σωστό είναι που η Κομισιόν, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Όλαφ προσπαθούν να ε, εποπτεύσουν το, όλο σύστημα. Θέλει να παρέμβει ο εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου πάνω σε αυτά που είπε η κυρία Γιάλασέντε. Ευχαριστώ την κυρία Γιάλα Σέντερ για την ερώτησή της. Φυσικά, εμείς έχουμε, κάνουμε τους ελέγχους μας με συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται και σημαντικά κονδύλια από πλευράς κρατών μελών ιδίως για την ε, συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών. Η Κομισιόν έχει συμφωνήσει με την έκθεσή μας και με τα μέτρα τα οποία προτείνουμε από πλευρά τεχνικού συνεδρίου. Σε αυτόν τον τομέα και στα πλαίσια του ελέγχου περιβαλλοντικών ε, ζητημάτων θα συντάξουμε μια έκθεση του χρόνου όπου ε, με θέμα, με θέμα συγκεκριμένο τη διαχείριση των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού το οποίο θα καλύπτει όλα τα θέματα της ε, ε, συλλογής, εναπόθεσης, διαχείρισης ε, και διάθεσης των λιμάτων στις εγκαταστάσεις. Όλη δηλαδή τη λειτουργία, η ζωή, η κλπ αυτή η έκθεση θα έχει οπωσδήποτε επιπτώσεις για τις μελλοντικές ελεγκτικές ενέργειες. Για τη σημασία του ρόλου του ελεγκτικού συνεδρίου θα ήθελα να σας πω ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα απάτης quello della Corte dei Conti è fondamentale anche per mettere in moto accertamenti poi sulle, sulle eventuali frodi. Do la parola all'onorevole διορθώθηκε ο έλεγχο, ε, χάρη σε εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Ο κ. Κλακάκης. Ρωτήσω τον εκπρόσωπο του ε, Court of Auditors εάν υπάρχουν δείκτες τους οποίους να χρησιμοποιούν ε, μεταξύ διαφορετικών χωρών ή στο σύνολο της κοινότητας, ειδικά σε ό,τι αφορά τον πιθανό υπερσχεδιασμό των έργων, δηλαδή έργα που καλύπτουν πολύ μεγαλύτερη ε, ε, που είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτό που πράγματι ανακαλύπτεται ότι ε, χρειάζεται και σχετικά με τις συγκριτικές δαπάνες μεταξύ των έργων στις χώρες της κοινότητας. Ευχαριστώ. Prego, Ε, ε, Πιστεύω ότι το ερώτημά σας είναι δύσκολο να απαντηθεί. Υπάρχουν προβλήματα όταν συγκρίνουμε παρόμοιες εγκαταστάσεις. Το έχουμε αντιμετωπίσει. Πώς δηλαδή ε, ξοδεύονται τα χρήματα για, τους, τη διαχείριση των λιμάτων. Είχαμε συντάξει, είχαμε προετοιμάσει ένα πολύ λεπτομερή έλεγχο. Όμως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κάθε φορά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη φάση του σχεδιασμού, διότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν παρεμβαίνει ούτε έχει καμία ευθύνη όταν σχεδιάζονται οι εγκαταστάσεις αυτές. Αυτή είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν η φάση σχεδιασμού και προετοιμασίας, διότι η Κομισιόν είναι και ο πρωταγωνιστής στη διαχείριση αυτών των πιστώσεων, μαζί με το, τα κράτη-μέλη βέβαια. Δεν έχουμε εμείς ένα σύστημα δικτών, διότι δεν έχουμε ε, δεν, είναι στον προγραμματισμό μας ε, να φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα δικτών, συγκριτικών δικτών. Η Κομισιόν είναι υπεύθυνη γι' αυτό. interventi? Άλλος κανείς? Ε, η κυρία Σέντερ. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι σοκαριστικό αλλά και ενδιαφέρον το ελεγκτικό συνέδριο φαίνεται να μας συστήνει και εγώ θα ήθελα να εμείνω και λίγο περισσότερο σε αυτό, διότι πρέπει να δούμε και μέχρι ε, ποιου σημαίου αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να είναι αποφασιστική σημασία σε αυτή η αλλαγή και στη λειτουργία των σταθμών βιολογικού καθαρισμού. Στη, σημεία 50 και 53 μας λέτε πού μπορούμε να εφαρμόσουμε την αρχή της μείωσης της ρήπανσης στην πηγή μέσω της μείωσης ή της πλήρους κατάργησης της χρήσης ε, απορριβατικών που περιέχουν ε, φωσφορικές ενώσεις. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ξεκινήσουμε δηλαδή από πλευράς Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία αναθεώρηση και να γίνουν λίγο πιο περιοριστικοί οι όροι για τη χρήση των φωσφορικών ενώσεων. Θέλετε να παρέμβετε. Στην έκθεσή μας, στο, στις παραγράφους 50 και 53, προτείνουμε, κάνουμε διάφορες προτάσεις, συστάσεις μάλλον, για την ε, χρήση απορριπαντικών ε, που περιέχουν ε, φωσφορούχες ουσίες. Και την... πρέπει να σας πω ότι συζητήσαμε ενδελεχώς μέσα στο ελεγκτικό συνέδριο και με, την, ε, με τους ελεγκτές μας το, τη μορφή αυτή των συστάσεων. Και έχουμε επίσης συζητήσει την διαδικασία που προτείνεται από την Κομισιόν. Και το συμπέρασμα αυτών όλων των συζητήσεων περιλαμβάνεται, έχει ασωματωθεί στην έκθεσή μας και δει στα συμπεράσματα. Δεδομένου ότι η Κομισιόν είναι ο διαχειριστής των ε, δημοσίων πιστώσεων, τα συμπεράσματά μας κατά τη γνώμη της Κομισιόν αρκούν για σωστή διαχείριση. Κύριος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε τρεις συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο από την ε, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και ένας από την Γενική Διεύθυνση Regio. Διαβάσαμε την έκθεση, την καλωσορίζουμε. Είχα τρία σημεία που είχα ετοιμάσει να αναφέρω, αλλά θα διεκπαιρεώσω και κάποια από τα σημεία που προέκυψα μετά από τη συζήτηση, εν συνεχεία. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ε, τις υποδομές που, χρήζονται με την, που χτίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Παραδείγματο χάρη τη σύνδεση των ε, αποχετεύσεων με τους βιολογικούς καθαρισμούς. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των επιχειρήσεων γενικά με βάση την νομοθεσία την, της πολιτικής συνοχής και των διαφορετικών ταμείων. Είναι μια πολιτική, ξέρετε πολύ καλά, που βρίσκεται σε εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 100 μελών ε, και περιφερειών. Και αυτό επηρεάζει τα πάντα. Είτε είναι νερό, είτε είναι απόβλητα, είτε είναι δρόμοι, είτε οτιδήποτε. Συγχρηματοδότηση δηλαδή. Σε πολλές περιπτώσεις ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε τα κράτη-μέλη ε, στο δικαστήριο και τα τέσσερα κράτη-μέλη που ελέγχονται τώρα για ανεπαρκή συλλογή ε, λιμάτων και για ανεπαρκή επεξεργασία των λιμάτων. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Το δεύτερο σημείο για την αναθεώρηση της οδηγίας για τον καθαρισμό της ηλίως αυτό είναι κατεπήγον, το ξέρουμε και η αξιολόγηση επιπτώσεων για αυτό που απαιτείται για τις νέες προτάσεις ε, είναι σε φάση σύνταξης και θα, είμαστε, θα είναι έτοιμη αυτή η αξιολόγηση στο τέλος του 2009, το τελευταίο τρίμηνο ή το αργότερο το πρώτο τρίμηνο του 2010. Και επομένως, ε, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ολοκληρώσει θα έχουμε ξεκινήσει μάλλον τη σύνταξη της νομοθετικής πρότασης, μπορεί και το πρώτο τρίμηνο του 2010. Τρίτον, σε ό,τι αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μην ξεχνάμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη βασική ευθύνη για την συλλογή, εφαρμογή και παρακολούθηση των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται. Γι' αυτό την ε, περίοδο προγραμματισμού 2007 με 2013 η Κομισιόν έχει απλουστεύσει την, το βασικό τρόπο εκτίμησης των προγραμμάτων. Μιλάμε για 25 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος. Και χωρίς τις ελάχιστες απαιτήσει, τα προγράμματα δεν υπάρχει περίπτωση να, να τα εγκρίνουμε για συγχρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για την στρατηγική διαχείριση της ηλίως και την διαχείριση και επεξεργασία των λιμάτων ε, από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτό Τώρα, τι σημαίνει. Ε, ακούσαμε αυτό που είπατε για το checklist, για τον κατάλογο και από τις αρχές του 2009 η Γενική Διεύθυνση Envy και ΡΕΤΖΙΟ ε, κατάρτισαν ένα τέτοιο κατάλογο για τα προγράμματα συγχρηματοδότησης κλιμάτων. για λίματα. Ε, στις 10 Ιουνίου συζητήσαμε την πρόταση αυτή με τα κράτη-μέλη και με τις αρμόδιες αρχές του Ταμείου Συνοχής. Επομένως, οι αρχές διαχείρισης, όλες οι συναρμόδιες αρχές είχαν τρεις μήνες να αντιδράσουν. Δεν ακούσαμε όμως καμία αντίδραση στις προτάσεις που τους κάναμε τότε, στις 10 Ιουνίου, και προτείνουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τελικά τον κατάλογο. Τώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, συζητήσεις που έγιναν για τις αλλαγές του Γενικού Κανονισμού της Πολιτικής Συνοχής, το κατόφλι για προγράμματα που θα ελέγχει η Κομισιόν, αν περάσει η πρόταση, θα αυξηθεί από 25 στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα συμπεριλαμβάνει δηλαδή και τα προγράμματα για το νερό. Επομένως, ο ρόλος των κρατών μελών τώρα σε αυτό το πλαίσιο επιμερισμένης ευθύνης και εταιρική σχέσης θα γίνει πολύ περισσότερο σημαντικό στο μέλλον από ό,τι είναι τώρα η Κομισιόν ζήτησε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να δίνουν πληροφορίες στις εκθέσεις εφαρμογής για τα προγράμματα που θα βρίσκονται μεταξύ 25 και 50 εκατομμύρια ευρώ και να δίνουν και λεπτομέρειες το των προγραμμάτων στις εθνικές ιστοσελίδες. Όπως κάνουμε και τώρα, θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε και περισσότερες επιτόπιες επισκέψεις στα κράτη-μέλη για να κοιτάξουμε αυτά τα προγράμματα τα οποία δεν θα κοιτάμε λόγω του, των τροποποίησεων στο, στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού. Τώρα, για τις ε, ερωτήσεις. Μίσης, ε, η κυρία Αγέλα Σάντες. Δεν υπάρχει αρκετή πραγμα, πραγματογνωμοσύνη. Σωστό, το αναγνωρίζουμε. Αλλά υπάρχει τεχνική αρρωγή ε, για τα Ταμεία Συνοχής και για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά αυτά τα προγράμματα. Και ακόμα και το, ταμείο, ε, το κοινωνικό ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση. Σε ό,τι αφορά το κόστος συντήρησης, ο κανονισμός με τις γενικές διατάξεις για, τις, για την πολιτική συνοχή έχει ειδικά άρθρα για την εφαρμογή της αρχής ορυπαίνων πληρώνει. Και χρησιμοποιούμε αυτά τα τέλη, ε, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα ε, του εκάστοτε υπεύθυνου να πληρώνει. Γιατί κάποιοι είναι πιο φτωχοί από άλλους. Επίσης προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2010, δηλαδη πρωτη 1η του 2011, να έχουν ένα πλαίσιο για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Και άλλος ένας τρόπος για να χρησιμοποιούμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτά τα τέλη. Επίσης, ο, κανονισμός, ο Γενικός Κανονισμός για τα Διαφορετικά Ταμεία προβλέπει πολύ καθαρά τη δυνατότητα οικονομικής διόρθωσης, εκεί που έχει γίνει υπερβολική επένδυση. Τώρα για τις φωσφορούχες και φωσφορικές ενώσεις, ε, θα δώσω το συνάδελφο, θα δώσω, θα το λόγο στη συνάδελφο. Thank you. Ε, ευχαριστώ. Όσον αφορά την ε, μετακίνηση την ε, προς ε, απορριπαντικά άνευ φωσφόρου η Κομισιόν έχει, κάνει, έχει συντάξει μια έξεση αξιολόγησης επιπτώσεων η ε, μετά από αυτή θα θα επακολουθήσουν διάφορες πρωτοβουλίες σε μεγάλο βαθμό ο φόσφορος και οι φωσφορικές ουσίες έχουν αφαιρεθεί από τα απορριπαντικά που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 66% μάλιστα των, ε, του πληθυσμού δεν χρησιμοποιεί πλέον ε, φωσφορούχα απορριπαντικά, με φόσφορο. Για στην, περιοχή της λεκάνης του Δούναβη όπου υπάρχει μία μονάδα διαχείρισης ε, ο φόσφορος θα αφαιρεθεί τελείως από τα οικιακά απορριπαντικά, τα απορριπαντικά δηλαδή για πλήση πλησίματος ε, μέχρι το 2015, 2010 με 2015. Υπάρχει αυτό το πενταετές πρόγραμμα δηλαδή για την απόρριψη, εξάλληψη τελείως ε, του περιεχομένου σε φόσφο σε όλα τα οικιακά απορριπαντικά πλησίματος ε, των χωρών που χρησιμοποιούν τη λεκάνη του Δούναβη. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς. Ε, σημείο 18. Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 4-2009. Η διαχείριση εκ μέρου τη Επιτροπή Συμμετοχή των Μη Κρατικών Φορέων στην Απτιαξιακή Συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο κύριο Στάι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου άρεσε αρκετά η έκθεση, αλλά συμφωνήσαμε με τον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου να κάνει αυτός πρώτα μια παρουσίαση και να πει τα βασικά στοιχεία και μετά να σας πω εγώ την απάντησή μου. Να δώσουμε λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Κίντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας δώσω μια εισαγωγή στη συζήτηση για την έκθεση αυτή. Το πρώτο σημείο ίσως που θα έπρεπε να επισημάνω είναι ότι η έκθεση αυτή ετοιμάστηκε προς το κοινό συμφέρον των δύο οργάνων μας, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιο συγκεκριμένα της Επιτροπής σας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι ε, η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού επανελειμμένως είχε ζητήσει από, την, ε, το Ελεγκτικό Συνεδρίο να συζητήσει το θέμα των μη κρατικών ε, φορέων στην αναπτυξιακή συνεργασία. Τώρα, υπάρχουν αρκετά έγγραφα τα οποία επισημαίνουν τη σημασία της ενίσχυσης της ε, συμμετοχής ε, και της συνεργασίας με τους μη κρατικούς φορείς ε, στην αναπτυξιακή συνεργασία τόσο στην ομοθεσία όσο και στα εσωτερικά έγγραφα της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως προς τη σημασία για τον προϋπολογισμό, η ροή κονδυλίων ε, τα οποία διοχετεύονται από μη κρατικού φορεί ε, στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι βάσει των στοιχείων που έχουμε για το 2007, τα οποία και χρησιμοποίησαμε, ε, είναι περίπου ένα δις ευρώ. Επομένως είναι πολύ σημαντικό το κονδύλιο ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου. Αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τρία βασικά ερωτήματα ελέγχου. Τα πρώτα δύο που αφορούν στο διτό ρόλο των μη κρατικών φορέων στο θέμα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Το πρώτο είναι πώς ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφάλισε ότι οι μη κρατικοί φορείς ε, συμμετέχουν αποτελεσματικά στην ε, διαδικασία της συνεργασίας, είτε ως εταίρος για τη δημιουργία στρατηγικών, και την εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής ε, στις χώρες ε, οι οποίες ευεργετούνται από το πρόγραμμα. Και το δεύτερο ερώτημα αφορούσε το ρόλο των μη κρατικών φορέων ως ε, ε εφαρμοστές των προγραμμάτων και εργολάβων των προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Ταμεία. Και το τρίτο ερώτημα σχετίζεται και με τα δύο προηγούμενα. Πώς ε, διασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, έχουν τις δυνατότητες οι μη κρατικοί φορείς να αυξήσουν τις δυνατότητες τους ε, να εφαρμόσουν καλά τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας και να είναι εταίροι τόσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και για τις κυβερνήσεις της ευεργετηθήσεις χώρες για τη μείωση της και την και την αύξηση της παραγωγής. Υπάρχουν αρκετέ λοιπόν παρατηρήσει και αρκετά ευρήματα τα οποία σχετίζονται και με τα τρία ερωτήματα. Θα μπορούσα αν θέλετε να σας τα συνοψίσω αναερώτηση. Πρέπει να πω ότι όλα όσα διαπιστώσαμε και όσα συστήνουμε έχουν ε, μεταφορθεί στο έγγραφο εργασίας που ετοίμασε ο κύριος Στά. Συμφωνούμε πλήρως με τα τελικά του συμπεράσματα. Είμαι στη διάθεσή σας λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Θέλετε να προχωρήσω και να τα παριθμίσω ένα προς ένα ή... και να σας πω τα βασικά συμπεράσματα του ελέγχου της έκθεσης ή θα τα κάνει αυτά ο εισηγητής. Είμαι στη διάθεσή σας λοιπόν για να απαντήσω ερωτήσεις για την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Στάι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κίνς και τους συνεργάτες τους για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν. Ακόμα και από τον ίδιο τον κλάδο ακούσαμε πολύ καλά νέα. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό το 2007. Μιλάμε για ένα 10% δηλαδή όλων των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται για την ανάπτυξη και την αναπτυξιακή συνεργασία. Κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι στη μετάφραση μιλάμε για φορείς, αλλά θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τη χρήση του όρου φορείς, διότι δεν μιλάμε μόνο για μη κυβερνητικές οργανώσεις, μιλάμε και για μη κρατικούς γενικότερα φορείς. Περιλαμβάνονται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όλοι όσοι συμμετέχουν στην ανάπτυξη, πολλές φορές έχουν και ε, ε εργάζονται υπό ευρωπαϊκή σκέψη και, ε, σκέπη συγγνώμη, και έλεγχο, αλλά υπάρχουν και ε, άλλοι φορείς, μπορεί να είναι ενώσεις ε, αγροτικές, θρησκευτικέ οργανώσεις, ε, εμπορικά επιμελητήρια, συνεταιρισμοί. Επομένως, στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αναφερόμαστε σε όλους όσους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ε, συμμετέχουν σε αυτό το κλάδο. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης ήρθα σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το λέμε πάντα, αλλά αυτή τη φορά είναι αλήθεια. Ήταν πολύ επικοδομητικές οι επαφές αυτές. Μίλησα με τον υπεύθυνο, με τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος είναι και εδώ σήμερα και ίσως ε, θα θέλει και να λάβει το λόγο αργότερα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου εξήγησε πώς βλέπει την κατάσταση και πώς ε, βλέπει τα όσα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προκειμένου να δοθούν κίνητρα ε, για τη συμμετοχή μη κρατικών φορέων στα αναπτυξιακά προγράμματα. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι αρχές είναι πάρα πολύ καλές και ε, Φαίνεται όμως ότι στην πράξη πόρο απέχουν αυτά που ελπίζουμε και φιλοδοξούμε από την πραγματικότητα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά ακόμα και έτσι φαίνεται να μην πηγαίνουν όλα καλά. Δεν ξέρω αν διαβάσατε την έκθεση αναλυτικά, να σας δώσω ένα παράδειγμα όμως. Το 2007 και το 2008 για τον προπολογισμό υπήρχε ένα κονδύλιο της τάξης των 380 εκατομμυρίων ευρώ. και υπήρχαν 4.400 τόσε αιτήσει. 380 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα έπρεπε να μοιραστούν σε αυτούς τους 4.400 ετούντες. Ζητούσαν λοιπόν χρηματοδότηση για προγράμματα τα οποία ήταν της τάξης περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη αδυναμία να δεχτούμε όλα τα προγράμματα. Έγινε μια πρώτη αξιολόγηση φυσικά ε, που σημαίνει ότι έγινε ένα ξεκαθάρισμα και φτάσαμε περίπου στις χίλιες αιτήσει. Μετά έγινε μια δεύτερη αξιολόγηση και ένα δεύτερο ξεκαθάρισμα και φτάσαμε περίπου στα 212 προγράμματα τα οποία είχαμε στον κατάλογο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, από τις 4.000 ε, τόσες έμεινε ένα 4,4%. Είναι πάρα πολύ ε, μικρό το ποσοστό και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε εμείς ως νομοθέτες και να σκεφτούμε και πώς μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε, να αναθεωρήσουμε τους κανονισμούς μας, τον εσωτερικό μας κανονισμό, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα προβλήματα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εχθέ μας διαβίβασε ε, τμήμα των εγγράφων τους, ε, στα οποία ε, καταδεικνύεται τι προσπάθειες έκαναν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου όσους συμμετέχουν στις αντιπροσωπείες να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι. Έγιναν πολλά σεμινάρια τα τελευταία χρόνια, σεμινάρια τα οποία διαρκούν αρκετές ημέρες και στην πρώτη μέρα του κάθε σεμιναρίου γίνεται μια απόπειρα να ενημερώσουμε το κοινό, γίνονται παρουσιάσεις σε PowerPoint, ε, εξηγούμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να προχωρήσουμε κλπ. Και μετά τη δεύτερη και την τρίτη μέρα των σεμιναρίων, Προσκαλούνται και εταίροι εκτός Ευρώπης ε, για να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα τα οποία μας έχουν ε, επισημάνει. ήρθαμε και σε επαφή με την οργάνωση Concord που είναι η οργάνωση ε, ομπρέλα των ευρωπαϊκών ε, μη κυβερνητικών φορέων που συμμετέχουν ε, στις διαδικασίες και ε, έτειναν ε, νου σε όλα τα αιτήματα, ε, στα όσα του ζήτησε το ελεγκτικό συνέδριο, ανέφεραν όλα τα προβλήματα και το ελεγκτικό συνέδριο οργανώθηκε πάρα πολύ καλά για την παρακολούθηση του θέματος αυτού και έγινε και μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων και γι' αυτό και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή. Από πλευράς μας και από πλευράς της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση αυτή λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη για τις επόμενες ημέρες έχει οργανωθεί και μία ακρόαση στην οποία θα είναι προσκεκλημένη η Concord ακριβώς για να ακούσουμε και τι ακριβώς συμβαίνει από τους ανθρώπους που εργάζονται επιτόπου στα προγράμματα. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πολύ καλά νέα. Αυτές όλες οι ε, διαδικασίες δεν θα πρέπει να μένουν μόνο στεγνά στον έλεγχο του προϋπολογισμού, αλλά θα μπορούν να ασχοληθούν και με τα θέματα αυτά και οι αρμόδιες ε, επιτροπές του Κοινοβουλίου. Εγώ βέβαια είμαι μέλος της Επιτροπής ε, Αναπτυξιακής Συνεργασίας, γι' αυτό ήθελα και να είμαι εισηγητή σε αυτή την έκθεση και έκανα μία απόπειρα στην έκθεσή μου να συνοψίσω όλα όσα έχουμε στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, ελπίζω να μπορέσετε να τα διαβάσετε αυτά που έγραψα και αυτό που προσπάθησα ήταν να μην συμπεριλάβω αποκλειστικά γενικές συστάσεις αλλά και κάποιες συστάσεις οι οποίες θα είναι πρακτικής φύσεως. Υπάρχουν και κάποιες προκλήσεις, προσκλήσεις όχι μόνο προς το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπάθησα να εστιάσω σε πολύ συγκεκριμένε λύσεις. Είναι αλήθεια ότι δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω τα πάντα, αλλά μία από τις συστάσεις που γίνεται είναι λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν προβλήματα στις αντιπροσωπείες επιτόπου που δεν έχουν αρκετές γνώσεις και αρκετή πείρα, γιατί να μην ε, κάνουμε μια απόπειρα κάποια στιγμή Παραδείγματο χάρη μέχρι το τέλος του 2010, σε όλες τις αντιπροσωπείες να υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος, ένα υπάλληλο Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα γνωρίζει όλα όσα χρειάζονται προκειμένου να συνδράμε αυτή την αντιπροσωπεία. Δεν ξέρω πώς να γίνει η διαμοσολάβηση για τα προγράμματα, πώς να γίνουν οι αιτήσει, πώς να υπάρχουν τα συνοδευτικά έγγραφα για τη χρηματοδότηση. Μιλάμε επίσης και για ανθρώπους που πρέπει να έχουν γνώσεις επιτόπου, για να μην υπάρχει και αυτό το πρόβλημα να ε, καθυστερούν οι διαδικασίες ακριβώς ε, λόγω έλλειψης γνώσεων. Αυτά λοιπόν είναι τα σχόλια τα οποία ήθελα να κάνω. Αυτό ήθελα να ε, σχολιάσω για την πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι ακόμα για το ελεγκτικό συνέδριο. Το να μπορούμε να υπολογίσουμε τα πράγματα έτσι, πατώντα ένα κουμπί σε έναν υπολογιστή και να λέμε ότι α, θα δώσουμε τα κονδύλια και μετά τα ξεχνάμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειαζόμαστε αξιόπιστα στοιχεία. Η Κομισιόν προσπάθησε να με εξηγήσει πώ ε, παρακολουθείται η όλη διαδικασία. και στις αρχές της διαδικασίας ε, διάθεσης των πόρων για το 2011 θα πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ε, ποια κονδύλια έφτασαν πού στον τομέα αυτό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε τα στοιχεία αυτά και για μας ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού να έχουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία όταν θα ετοιμάσουμε τον προπολογισμό για το 2011. Κάτι ακόμα. Θεώρησε ότι ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή πλέον να σκεφτούμε καλά όλο αυτό το θέμα της συγχρηματοδότησης. Ε, πώς μπορούμε να το αναθεωρήσουμε προκειμένου οι οργανώσεις, τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι οργανώσεις τρίτων χωρών του Νότου, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ταμεία και να έχουν ε, μια διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία, να ξέρουν ε, πώς πάνε τα πράγματα. ώστε όταν θα τεθεί θέμα αναθεώρησης του χρηματοοικονομικού στοιχείου θα πρέπει να έχουμε και τη χρηματοοικονομική αναθεώρηση για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη και κάποια σημεία, κάποιους προβληματισμούς ε, που διαπιστώσαμε στην ε, έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και όχι απλά να τα αναφέρουμε επιγραμματικά, αλλά να αναγνωρίζουμε ότι ως συνομοθέτες έχουμε και εμείς ευθύνη. Διαπίστωσα επίσης ότι ε, πέραν της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου υπάρχει και μια σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνεργασία ε, την αναπτυξιακή. Έχω τα στοιχεία για το έγγραφο, έχω και τη διεύθυνση την ηλεκτρονική στην οποία μπορείτε να βρείτε το έγγραφο. Θεωρώ ότι το να διαβιβάζονται τέτοια έγγραφα είναι πολύ σημαντικό για να καταλήξετε σε συμπεράσματα για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είμαι στη διάθεσή σας αν οι συνάδελφοι ή το ελεκτικό συνέδριο έχουν ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέμπερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι η Κομισιόν συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό τις παρατηρήσεις του εισηγητή και του ελεγκτικού συνεδρίου. Το πρόβλημα το οποίο αναφέρεται σε αυτή την έκθεση είναι περίπλοκη, περίπλοκο, πρέπει να το σκεφτούμε από κοινού, πρέπει να συνδιαλλαγούμε, ούτως ώστε να δούμε τι ιδέες έχει ο καθόνας. Η ακρόαση που θα γίνει τη Δευτέρα είναι ευπρόσδεκτη γιατί ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικός διάλογος. Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί με δεκάδες, ε, κατοντάδες, χιλιάδες οργανώσεις της κοινωνίας ε, των πολιτών. Μιλάμε για κοινωνίες των πολιτών σε 150 χώρες. Έτσι. Ε, είναι μια πρόκληση και όλες οι καλές ιδέες είναι ευπρόσδεκτες. Ελπίζω να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από συζητήσεις με όλους. Ε, από τους ενδιαφερόμενους φορείς, δηλαδή τους μη ε, κρατικούς φορείς, τους ε, Ευρωπαίους, αλλά και τους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις τρίτες χώρες. Το Κοινοβούλιο, το Ελεκτικό Συνέδριο και την Κομισιόν. Με αυτόν τον τρόπο, νομίζω, με τέτοια σύνθεση θα φτιάξουμε ιδέες πιο, και προϊόντα πιο προσαρμοσμένα στα προβλήματα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, να σταθώ σε κάποια σημεία του που ανέφερε ο κύριος Στάις, να έχουμε σε κάθε αντιπροσωπεία ειδικού για τα προβλήματα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ναι. Φυσικά όμως πρέπει να τονίσω ότι αυτή η απάντηση έχει κάποιους περιορισμούς. Και οι περιορισμοί αυτοί είναι οι ανθρώπινοι πόροι. Η Κομισιόν δεν μπορεί να αποφασίσει, δεν είναι ρόλος της, μπορεί να το ζητήσει, αλλά οι ανθρώπινοι πόροι είναι η δημοσιονομική αρχή που τους διαθέτει. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ λοιπόν ότι θα διαθέσουμε τις, τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους. Φυσικά θα πρέπει να διχειριστούμε το σύνολο της συνεργασίας. Ε, συνεργασία με τους μη κυβερνητικού φορείς είναι πολύ σημαντική. Είναι της τάξης του 10% αυτού που ξοδεύουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αλλά υπάρχει και ένα 90% δίπλα που πηγαίνει σε άλλα προγράμματα, σε άλλα project, σε άλλα σχέδια και όλα θα πρέπει αυτά να τα διαχειριστούμε. Ο στόχος μας είναι φυσικά να έχουμε ειδικού παντού, στο βαθμό του δυνατού πάντα. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, τη δυνατότητα να μας στάνουν δεδομένα ε, ώστε να το πιο ακριβή και πιο πλήρη. Αυτό το πρόβλημα το βλέπουμε παντού. Στις διεθνείς οργανώσεις, το, στο, στους, μη στους μη κρατικούς φορείς, ε, σε όλα τα επίπεδα υπάρχει και τίθεται αυτό το πρόβλημα. Οπουδήποτε υπάρχουν κοινοτικέ δαπάνε. Φυσικά είμαστε έτοιμοι να βελτιώσουμε τα πράγματα, κάνουμε τέτοιες προσπάθειες. Μπορούμε να το δούμε αυτό στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2011 και ούτως ή έχουμε κάνει ήδη προσπάθειες. Ε, γιατί έχουμε υλοποιήσει προγράμματα που επιτρέπουν στους μη κρατικούς φορείς να καταχωρηθούν. Γιατί πρόβλημα, υπάρχει και πρόβλημα όγκου δεδομένων. Όταν έχουμε να κάνουμε τόσους πολυάριθμους φορείς, υπάρχει δυνατότητα όγκου δεδομένων και διαχείρισή τους. Να τονίσω και ένα θέμα που έχει να κάνει με τη, με τη σύνεση. Και τα καλύτερα μηχανοργανωμένα συστήματα μπορούν να φτάσουν σε ένα επίπεδο. Δεν μπορούμε να του ζητάμε κάθε μέρα διαφορετικά δεδομένα. Ό,τι και να ζητάμε εξαρτώνται από την εισαγωγή των δεδομένων, την καταχώρηση των δεδομένων. Και η εισαγωγή περνάει από του ανθρώπου. Και οτιδήποτε περνάει από του ανθρώπου είναι περιορισμένο. Κάθε μέρα μα ζητάνε να συμπληρώσουμε μηχανοργανωμένα συστήματα με δεδομένα και παραμέτρους που αλλάζουν κάθε μέρα. Παραδείγματο χάρη, τη μία μέρα θέλουν να βάλουμε και να επικαιροποιήσουμε ξέρω εγώ, τον αριθμό των χιλιόμετρων ε, δρόμων που φτιάξαμε ή τους τόνους ε, ασφάλτου που ρίξαμε κτλ. Σας παρακαλώ λοιπόν όλους, ελεγκτικό συνέδριο, κοινοβούλιο, να μας συμπονέσει, να καταλάβει το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι και ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε περιορισμένα πράγματα. Δεν μπορούμε με, με σε μία στιγμή, ε, μία νυχτή να τα ρυθμίσουμε όλα. Χρειάζεται χρόνος για το σύστημα της συγχρηματοδότησης. Συμφωνώ απόλυτα. Και εξάλλου στον οικονομικό κανονισμό έχουμε οι δυνατότητες χρηματοδότησης 100% σε κατεπίγουσες περιπτώσεις. Τούτου λεχθέντος, με κάθε σεβασμό, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η απέτηση συγχρηματοδότησης είναι μια απέτηση που την θέλατε κι εσείς, τη θέσατε κι εσείς στο παρελθόν. Και αν μπορώ να κάνω και ένα προσωπικό σχόλιο, νομίζω ότι έχει μια δικαιολογία απόλυτα σωστή. Ε, διαχειριζόμαστε πολύ καλύτερα τα χρήματα και τα προγράμματα όταν συμμετέχουμε και εμείς οι ίδιοι, παρά όταν μας τα δίνουν απλώς από αλλού. Είναι θέμα ιδιοκτησίας των πόρων. Επίσης, και δεν υπάρχει κανένας λόγος οι, κρατικοί, μη κρατικοί φορείς να μην συνεισφέρουν και αυτοί με ένα περιορισμένο τουλάχιστον τρόπο. Ναι, σε ορισμένα προγράμματα ναι, να υπάρξει 100% ε, χρηματοδότηση όταν υπάρχει, υπάρχουν κρίσιμες και πήγουσες ανάγκες, αλλά το να το κάνουμε αυτό συστηματικά, ε, προσοχή. Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία που ήθελα να σχολιάσω. Επαναλαμβάνω, είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε με εσά, με το Ελεκτικό Συνέδριο, με την Επιτροπή σας και με την Επιτροπή Ανάπτυξης για να βελτιώσουμε όσο μπορούμε, έστω και λίγο, το αποτέλεσμα των εργασιών μας γύρω από, τις μη, από τους μη κρατικούς φορείς, λαμβάνοντας υπόψη ότι, έχουμε, ότι παίζουμε σε πάρα πολλά ταμπλό, σε 150 ή 200 χώρες, ε, ότι οι χώρες αυτές είναι κυρίαρχες, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και έχουμε να κάνουμε και μια πλειάδα τέτοιων φορέων. Επομένως, θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να τα λάβουμε υπόψη μας για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριος Μπέρμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω μετά τη θαυμάσια παρουσίαση του κυρίου Στάς. πιστεύω ότι αυτό που κάνατε ήταν απολύτως απαραίτητο, αυτό χρειαζόταν δηλαδή και συντοψίσατε πολύ καλά την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για μη κρατικού φορείς και την ε, συμβολή τους, την εμπλοκή τους σε προγράμματα ανάπτυξης. Κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με μη κρατικού φορείς, παραπονιούνται ότι δεν τους επιτρέπουν να συμμετάσχουν όσο θα ήθελαν, ότι οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ περίπλοκες κάθε φορά που πρέπει να παρουσιάσουν προτάσεις και ότι οι διαδικασίες εποπτείας και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων τους που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται ικανοποιητικά, δεν γίνεται σωστά. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε πλέον την εξουσία να αξιολογήσουμε την πολιτική της Κομισιόν και είναι πολύ σημαντικό σημείο αυτό και όσον αφορά την Επιτροπή Ανάπτυξης. Έχουμε ε, πολλούς φακέλους ε, για όλες τις χώρες όπου η Κομισιόν ε, προσφέρει, δίνει αναπτυξιακή βοήθεια και στην προηγούμενη θητεία είχα ε, συζητήσεις, ε, σοβαρές συζητήσεις κάνει με την Κομισιόν σε αυτά τα αναπτυξιακά θέματα και για τα προγράμματά τους παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο η Κομισιόν μέσω αυτών των αναπτυξιακών προγραμμάτων για την κοινωνική συνοχή. Όταν εφαρμόζονται αυτά τα προγράμματα έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις κοινωνίες. Το καθεστώς της ιδιοκτησίας, ownership, ιδιοκτησία, ε, ε, είναι μια λέξη πολύ της μόδας. Δεν είναι πολύ κομψή η ορολογία αυτή, αλλά πιστεύω σε αυτό το πλαίσιο είναι σωστή και οι επικρίσεις που παρουσιάζονται στην έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου είναι σαφέστατες. Μπορούμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις επικρίσεις, αυτή την κριτική, σαν ε, οδηγό για να αναθεωρήσουμε την πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας από την πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πιστεύω ότι αυτό θα το κάνουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευτυχής που η έκθεση αυτή δημοσιεύτηκε και αφορά τη δράση μη κρατικών φορέων στον τρίτο κόσμο. Υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ δεσμεύσεων και εφαρμογών, δηλαδή δεσμεύσεων, ε, προτάσεων που έχουν γίνει εγγράφος ε, και δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί και του τι έχει συμβεί πραγματικότητα. Με την αναπτυξιακή βοήθεια τώρα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα, μια, ένα καθεστώς μικροδιαχείρισης για να βελτιώσουμε την κατάσταση σε αδύναμες ε, περιοχές, σε μη ανεπτυγμένες περιοχές. Οι πιστώσεις αυτές μέσω της Κομισιόν ε, διοχετεύονται σε πάρα πολλές ε, περιοχές του τριτού κόσμου και βλέπουμε εδώ ότι πολλές φορές αυτές οι πιστώσεις, αυτή η αναπτυξιακή βοήθεια δεν λειτουργεί. Δεν δουλεύει το σύστημα. Πρέπει λοιπόν ε, να σώσουμε ό,τι μπορούμε η έξεση αυτή προτείνει περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη στελέχη για την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά εγώ νομίζω το πρόγραμμα είναι βασίτερο. Εάν θέλουμε να γίνει σωστή εφαρμογή της αναπτυξιακής βοήθειας και γενικά της αναπτυξιακής πολιτικής, θα, πρέπει να, έχουμε μία, να κλείσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ λέξεων και πράξεων. Όπου θέλουμε να λειτουργήσει σωστά δεν λειτουργεί και όπου δεν, ε, δεν χρειάζεται εκεί λειτουργεί. Λοιπόν, ε, ένα μέλος των Πρασίνων έχει παρουσιάσει αυτή την έκθεση και την υποστηρίζει και η σοσιαλιστική ομάδα. Θα γίνει μία ακρόαση και θα ήθελα να είμαι παρόν στην ακρόαση αυτή ε, εκτός αν δεν με καλέσουν βέβαια, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε πιο κριτικά, πιο προσεκτικά το ρόλο των ε, μη κρατικών των φορέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και να δούμε πώς ε, δρούν ε, στον τρίτο κόσμο. Ενεργούν πραγματικά προς το συμφέρον των πληθυσμών εκεί ή προς το δικό τους συμφέρον, προς το ίδιο συμφέρον δεν αρκεί το να μπορούμε να σώσουμε ό,τι έχει απομείνει για σώσιμο. Πρέπει να προχωρήσουμε πέραν αυτού. Ο εκπρόσωπο του ελληνικού Συνεδρίου θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με, θα ήθελα να κάνω μερικά, μερικές τελικές παρατηρήσεις μετά από αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση η Κομισιόν έχει δηλώσει ότι η έκθεσή μας είναι λίαν ε, ισόρροπη, ότι παρουσιάζει όλα και έχει εντοπίσει όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν πολλά προκλήσεις ε, τις οποίες πρέπει να εντοπίσει η Κομισιόν και τα γνωρίζει. Εμείς αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχει κάνει η Κομισιόν μετά από την βάση της εκθέσεως μας αυτή και θα κάνει και στο μέλλον. Δεύτερον, ε, εξ αρχής γνωρίζαμε την ε, αξιολόγηση της ίδιας της Κομισιόν για την αναπτυξιακή βοήθεια και την ε, δράση των μη κρατικών φορέων. Πάντοτε λοιπόν διαβάζουμε και άλλες εκθέσεις από διαφορετικές πηγές ή όπου τέλο πάντων έχει γίνει μια άλλη αξιολόγηση, μια εργασία, μια μελέτη που μπορεί να βοηθήσει τη δική μας έκθεση. Σε αυτή την ειδική έκθεση αναγνωρίζουμε ότι η, τα κριτήρια αναφοράς για το πλαίσιο αξιολόγησης της Κομισιόν δεν είναι ακριβώς αυτά που θα επιθυμούσαμε, τόσο σαφή δηλαδή και συγκεκριμένα. Εν πάση περιπτώσει, η Κομισιόν έχει δεχθεί ότι θα πρέπει να βελτιώσει ε, την εποπτεία της φάσης σχεδιασμού στις ε, ωφελούμενες χώρες των διαφόρων προγραμμάτων και την αύξηση και βέλτιστη χρησιμοποίηση του δυναμικού των έργων. Τη Δευτέρα απόγευμα στα, στην ανοιχτή ακρόση πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την παρουσία όλων των ενδιαφερομένων διότι εκεί θα ακουστούν διάφορες προτάσεις ε, για τη μελλοντική πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. και ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Μία-δύο αντιδράσεις. Καταρχάς τόσα είπε ο κύριο Βέμπερ και εν συνεχεία τόσα είπε ο κύριο Έπινγκ. Ο κύριο Βέμπερ μίλησε για αυτό που ανέφερα στην έκθεσή μου για την ε, συγχρηματοδότηση και την χρηματοδότηση 100%. Συμφωνώ με αυτό που είπε. Δεν θεωρώ ότι κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να χρηματοδοτείται κατά 100%. Απλώς θα πρέπει να αφήνεται η δυνατότητα. Γιατί σε μερικές περιπτώσεις είναι πραγματικά καλή ιδέα και είναι πολύ καλύτερα να υπάρχει χρηματοδότηση 100% παρά συγχρηματοδότηση από διάφορους ε, χρηματοδότες. Αν υπήρχε εξάλλου χρηματοδότηση 100% όλων των προγραμμάτων των μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων, δεν θα ήταν πια μη κυβερνητικέ οργανώσει. Θα και, πρέπει και οι ίδιε να εξακολουθήσουν να κάνουν προσπάθειε για να βρίσκουν τουλάχιστον ένα τμήμα των κονδυλίων που του χρειάζονται για τη λειτουργία του. Τώρα, για αυτά που είπε ο κύριο Σέπινγκ. Κατανοώ τι ε, ιδεολογικέ σα απόψει για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι κλασική νεοφιλελεύθερη και άκρος, μάλιστα νεοφιλελεύθερη, άποψη αυτή. Αναφέρατε τον προηγούμενο εργοδότη σας, τον κύριο Μπόλκενστάιν. Ε, δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ και απόλυτα μαζί του. Νομίζω ότι οι μη κυβερνητικοί και μη κρατικοί φορείς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Φέρνουν αποτελέσματα. Δεν ε, φέρνουν αποτελέσματα 100% πάντα, αλλά έτσι συμβαίνει αυτό. Αυτή είναι η ζωή. Επίσης, ε, είσαστε ευπρόσδεκτοι, κυρία μου, στην ε, ακρόαση που θα κάνουμε. Εξάλλου, όλοι οι βουλευτές είναι πάντα ευπρόσδεκτοι σε όλες τις ακροάσεις και μάλιστα περιμένουν με υπομονησία να γίνει αυτή η ακρόαση και η συζήτηση στα πλαίσια της ακρόασης. Ευχαριστώ, κύριε Στάες. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Όχι. Πάμε στην τελευταία έκθεση για τη διαχείριση στη φάση ανάπτυξη, ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διαχείριση στη φάση ανάπτυξης και επιβεβαίωση του προγράμματος Γκαλιλαίο. Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με το πρόγραμμα Γκαλιλαίου ετοιμάζουμε ένα ευρωπαϊκό δορυφορικό πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ευρεία ακτίνα και όσον αφορά το FES σύστημα μεταφορών. Η έκθεση που μας έδωσε το ελεγκτικό συνέδριο είναι σαφώς ε, σημαντική έγκαιρη, πολύ καλά διατυπωμένη και απαραίτητη σε εμά όλους. Για ποιο λόγο. Διότι το σύστημα στη φάση ανάπτυξής του και ε, ε, επικύρωσής του προέβλεπε ένα πάγιο ποσό το οποίο θα έπρεπε να ε, χρησιμοποιηθεί από το 2001 έως το 2005. Έπρεπε να εκταμιευθούν 1,1 δις ευρώ από, το, από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το 76% έπρεπε να καλυφθεί από ιδιωτικά κεφάλαια. Έχουμε λοιπόν την εξής κατάσταση. Το κόστος διπλασιάστηκε, δεν θα κοστίσει 1,1 δις ευρώ το πρόγραμμα, αλλά πάνω των 2, 2 δις ευρώ και οι εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν το 2005. Κατά πάσα πιθανότητα θα ολοκληρωθούν το 2010 και δεν θα υπάρχει συγχρηματοδότηση κατά 1 τρίτο από δημόσια ταμεία, αλλά κατά 100% και τα 3 τρίτα δηλαδή. Τι με λιγενέστε. Υπήρχαν 33 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ για την εμπορική φάση, η οποία υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πέρσι, αλλά η εμπορική φάση θα ολοκληρωθεί το 2014 και δεν θα έχουμε 3,3 δις ευρώ, αλλά θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα 6 δις ευρώ. Και η συμμετοχή δημοσίων κονδυλίων δεν θα είναι 33% αλλά και πάλι κατά πάσα πιθανότητα κατά 100%. Επομένως, ε, η έκθεση αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και η ανάλυση των αιτίων που μας οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση. Οι παράγοντες αυτοί, οι οποίοι αξιολογήθηκαν από το ελεκτικό. συνέδριο μπορούν να αξιολογηθούν ως εξή. Καταρχάς υπήρχε κακοδιαχείριση του προγράμματος Γαλιλαίο τόσο στη φάση ανάπτυξής του όσο και στη φάση επιβεβαίωσης. Και δεν ξέρουμε και πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα δεν καθορίστηκε σταφώς ο ρόλος των ε, ε, βασικών διαμεσολαβητών. Ο αρχικός φορέας ήταν η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία η οποία ήταν υπεύθυνη για τα τεχνικά θέματα και τα θέματα περιεχομένου του προγράμματος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν υπεύθυνη για τον καθορισμό των στόχων, για τον καθορισμό των πολιτικών και την ε, διαδικασία των επενδύσεων. Τι πήγε στραβά τώρα. Όλα πήγαν στραβά κατά ε, το νόμο του Μέρφυ, άλλωστε. Η δημόσια ιδιωτική εταιρική σχέση, για παράδειγμα, δεν ήταν πολύ καλά καθορισμένοι κανόνες, ε, οι εταίροι οι ιδιωτικοί δεν ε, συμμετείχαν τελικά γιατί ο δημόσιος φορέας δεν ήταν έτοιμος να δεχτεί ιδιωτική, ιδιωτικούς φορείς και για το λόγο αυτό υπήρχε χρηματοδότηση Καταλήξαμε μάλλον στη χρηματοδότηση του 100%. Ε, υπερβήκαμε το κόστος, ε, δεν τηρήθηκαν οι προσθεσμίες, ε, οι διαχειριστές του προγράμματος δεν ήταν έτοιμοι από πλευράς ουσίας και περιεχομένου και δεν υπήρχε και ένα μακροπρόθεσμο όρομα για την καθοδήγηση, για τη διαχείριση ενός προγράμματος αυτής της ε, μορφής. Επίσης, δεν έγιναν διαπραγματεύσεις για την εκχώρηση με κατάλληλο τρόπο. Αυτές αν θέλετε είναι ευθύνε Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία δεν κατάρθωσε να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο της διαχείρισης ε, όλου του προγράμματος. Έχουμε επίσης και τις δραστηριότητες των κρατών μελών και εδώ συμφωνώ με το ελεκτικό συνέδριο ότι υπάρχει μία σειρά από παρεμβάσεις των κρατών μελών στον τομέα αυτό που οφείλονται στο γεγονός ότι όλες αυτές οι χώρες μέλη ήθελαν να προασπίσουν τα συμφέροντα της δικής τους ε, διαστημικής διάστασης, τα οικονομικά τους συμφέροντα στις διάφορους ε, μειοδοτικούς διαγωνισμούς και υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέδειξε ιδιαίτερη αδυναμία και δεν αντιτάχθηκε σε αυτή την τάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε σε αυτές τις ε, αντιρρήσεις και τις ενστάσεις, αλλά είναι η παραδοσιακή απάντηση, γιατί είναι η συνήθις απάντηση που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει ότι υπάρχουν προβλήματα, λέει ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν στο μέλλον, αυτά λέει η Επιτροπή. Και επειδή υπάρχουν προβλήματα, συστήσαμε και μία ειδική ομάδα και ίσως με αυτό το, την ειδική ομάδα να λύσουμε και τα προβλήματά μας. πήρα το θάρρος να παρουσιάσω και κάποιες συστάσεις ε, προς το Ελεκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη μου σύσταση είναι ότι ε, είναι πονίδιστη αυτή η καθυστέρηση των πέντε ετών και προτείνω να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει σαφώς βάσει των ε, ε, τρεχουσών προθεσμιών με πέντε χρόνια ήδη καθυστέρησης τα πιο βασικά πολιτικά σημεία ε, και τους πολιτικούς στόχους αυτού του συστήματος. Πρέπει να καθορίσει ποιοι είναι οι λειτουργικοί στόχοι και ποιος είναι και ο χάρτης πορείας ο οποίος θα μας οδηγήσει στην πλήρη λειτουργία, εμπορική λειτουργία του συστήματος. Προτείνω επίσης να εκφράσουμε την ανησυχία μας, διότι αυτό το κοινό εγχείρημα, τον Γαλιλαίο, δεν ε, επέτυχε τους στόχους που είχαμε καθορίσει. Και λόγω της ε, δομής διαχείρισης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δεν διασφάλισε σε καμία περίπτωση επιτυχία. Τρίτον, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όσοι συνεισφέρουν θα πρέπει να ενημερώνονται για τα όσα συμβαίνουν και το πώς χρησιμοποιούνται οι χρηματοδοτήσεις για αυτό το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Επίσης θα πρέπει να διευκρινίσουμε ποιοι είναι οι πολιτικοί λόγοι που επισέρχονται. Πώς μπορούμε να πούμε ότι εμείς αφενός θέλουμε να υποκαταστήσουμε το αμερικανικό σύστημα και να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα και το ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς τεχνολογικής σε μεγάλο βαθμό να βασίζεται σε συστήματα και στοιχεία τα οποία δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή έχουμε υπερβεί το κόστος κατά 100%, ε, έχει παραταθεί η διάρκεια κατά 100% σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα. Ποια είναι η μελέτη κόστος-όφελος σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα το οποίο είχαμε συζητήσει πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια άλλωστε. Τι ακριβώς θα είναι αυτό το καλλιλέο, σε τι θα μετατραπεί. Να περάσω τώρα στις ευχαριστίες. Ευχαριστώ το ελεκτικό συνέδριο, τον πρόεδρο και όλους τους συναδέλφους για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο λόγος στο ελεκτικό συνέδριο, η κυρία Κέρστη Κάλιουραϊτ. Thank you, Chairman. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά τον ε, κύριο Λιμπερότσκι και διάβασα και την έκθεση που προετοίμασε και σαφώς ε, αντανακλά τα σχόλια της έκθεσης του, Ευρωπαϊκού, του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Γαλιλαίο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τόσο ευρία αξιολόγηση και ένας τόσο μεγάλος έλεγχος σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και είναι κατανοητό ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σημειώθηκαν διάφορες αλλαγές και διάφορα άγνωστα στοιχεία. Προσπαθήσαμε να αποκαλύψουμε αυτά τα άγνωστα στοιχεία και για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ε, στο Κοκομπού μία περιστατωμένη έκθεση. Και τι έγινε επιτέλους με αυτό το Γαλιλαίο, διότι όταν αρχίσαμε την ε, έρευνα και τη μελέτη μας, πολλά πράγματα ε, είχαν ήδη εντοπιστεί. Πιστεύω ότι με τις συστάσεις που κάνουμε θα βοηθήσουμε όχι μόνο την επιβίωση του Γαλιλαίου, αλλά και όλους τους άλλους σχεδιαστές ε, και αξιολογητές και ελεγκτές των κοινών προγραμμάτων να εκτελέσουν καλύτερα τις εργασίες τους και να λειτουργήσουν καλύτερα τα κοινά προγράμματα του μέλλοντος. Η κυρία Γιάλας, ο κύριος Οντή πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον εισηγητή μας για τη δουλειά του και να πω στο ελεκτικό συνέδριο ότι αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και είναι πολύ χρήσιμο να βλέπουμε πώς πάει μια διαδικασία, για την οποία εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε βέβαια περήφανοι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε πού φτάσαμε. Γιατί τα είχαμε μπλέξει εντελώ. Δεν καταλαβαίναμε πού ήμασταν. Και νομίζω ότι αυτή η έκθεση ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Καταρχά, θέλω να πω ότι είμαι λιγότερο αυστηρό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον συνάδελφο. Γιατί αν απέτυχε στην πρώτη φάση αυτό το θέμα, προσωπικά πιστεύω ότι απέτυχε βασικά όχι η Κομισιόν, αλλά ο ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικό τομέα δεν τα κατάφερε με διάφορες πολιτικές επιπτώσεις, έτσι, προφανώς. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι διδαχθήκαμε για τις μεγάλες υποδομές. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γνώρισαμε κάποιες ε, δυσκολίες. Παραδείγματο χάρη ε, το τούνελ της μάχης. Και χαιρετίζω την προσπάθεια του Ζακ Μπαρό και όλου του Κοινοβουλίου που ζήτησε να επανέλθουν αυτά τα προγράμματα στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί ήταν ο μοναδικός τρόπος για να βγούμε με το κεφάλι ψηλά και περήφανοι από αυτόν τον κικαιώνα. Λίγο εκτός θέματος είμαστε. Ίσως να μιλήσω λίγο για τα λογιστικά του προγράμματος. Γιατί όταν μιλάμε για τη συγγραφή υποχρεώσεων με την, ε, και το συζητάμε με την Κομισιόν, μιλάμε και για τους ε, ενοποιημένους ε, λογαριασμούς, αλλά και για τους, το μέλλον. Για το 2007 είχαμε ψηφίσει ένα ερωτηματικό. Καταρχάς, ρωτήσαμε σε ποιον ανήκει το Γαλιλαίο σήμερα. Πώς μπαίνει το πρόγραμμα Γαλιλαίο στου ενωπημένου ε, λογαριασμούς. Δεν είχε γίνει στις 31 Δεκεμβρίου του 2007 αυτό. Δεν είχε μπει το Γαλιλαίο. Ε, θα κοιτάξω και του λογαριασμού το 2008. Ε, δεν έχω προλάβει να το κοιτάξω ακόμα. Το θέμα είναι πώς θα μπουν στους λογαριασμούς τα έξοδα για το Γαλιλαίο. Ε, κύριε Πρόεδρε, Καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον συνάδελφο τον κύριο Λιμπεράσκη για την ε, πολύ σημαντική μελέτη που έκανε, κυρίως για τα συμπεράσματα και τις συστάσεις και επίσης και το ελεγκτικό συνέδριο για την πολύ πλήρη έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας δίνει τη ευκαιρία να μελετήσουμε εις βάθος ε, τα προβλήματα του Γαλιλαίου και να προσπαθήσουμε προληπτικά τουλάχιστον να μην επαναληφθούν αυτά σε κάποιες περιπτώσεις στη νέα περίοδο του Γαλιλαίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί το ίδιο έκανε και ο κύριος Σοντή. Μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα του οποίου τη διαχείριση έχει Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ουσιαστικά η διαχείριση είναι και διακυβερνητική και ε, υπάρχει και ο κίνδυνος να την περάσουμε στον ιδιωτικό τομέα η οποία έχει και τους ευθύνες του και δεν μπορεί να προχωρήσει κάποια πράγματα. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο, δεδομένου ότι αναλύει πάρα πολύ καλά πώς μπορεί ένας ιδιωτικό, μια ιδιωτική σύμπραξη με το δημόσιο μπορεί να καταλήξει μια τέτοια αποτυχία και μας δίνει και όλα τα στοιχεία. Αλλά θα ήθελα να δω αν μπορείτε να εμβαθύνετε λίγο περισσότερο και εγώ υποστηρίζω και εδώ ένα από τα συμπεράσματα του εισηγητή με μεγάλο ενθουσιασμό να ζητήσουμε από το ελεκτικό συνέδριο να κάνει μια νέα μελέτη για το διάστημα από το 2000 έως το 2006 διότι από αυτή την εξαιρετική έκθεση μπορούμε να αποφύγουμε κάποια σκακοτοπιές οι οποίε ε, μπορεί να επανελευθούν, να υπάρχουν, ελοχεύει κίνδυνο να έχουμε εκ νέου τέτοια προβλήματα. Θα θέλαμε λοιπόν να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο πώς ήταν ο ρόλος του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, διότι από εκεί θα μάθουμε πάρα πολλά και ε, θα δούμε και τι μπορεί να γίνει σε μελλοντικέ ε, συμπράξει τέτοιε που προσπαθούμε να κάνουμε. Επίσης, το αναλύσαμε, ήταν αποτυχία, δεν τίθεται θέμα εδώ, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό θέμα το οποίο άπτεται του Γαλιλαίου αλλά και άλλων ε, ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποδομών που είναι το γεγονός ότι έχουμε πολιετή προγραμματισμό στον προϋπολογισμό. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους, κυρίως για τον ιδιωτικό τομέα, ήταν να προβλέψουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση πέραν των ε, κοινοτικών προϋπολογισμών. Τώρα όμως που είναι 100% δημόσια χρηματοδότηση υπάρχει αυτή η πτυχή. Πώς μπορούν λοιπόν αυτά τα προγράμματα, πολλές φορές τα ζητάω αυτά από το ελεγκτικό συνέδριο, θα ήθελα να μου απαντήσουν, με ποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε κυρίως την αξιολόγηση και την πρόβλεψη ε, για τους κινδύνους σε προγράμματα αυτή τη μορφή που έχουν πολυετή προπολογισμό, ο οποίο πηγαίνει πέραν των δημοσιονομικών προεκτικών. Και επίση θα ήθελα να επαναλάβω το αίτημα να έχουμε μια νέα έκθεση από το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν ξέρω πώς είστε από προσωπικό και από αυτός εργασία, αλλά εμένα μου φαίνεται ότι είναι κατεπήγον αυτό, διότι από εκθέσει που έχουμε λάβει διαπιστώνω ότι οι νέε συζητήσει με τα κράτη-μέλη δείχνουν ότι ένα μέρος της συντήρησης του έργου θα γίνεται και πάλι με σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Θα ήθελα λίγο λοιπόν να δω τι γίνεται με αυτό το νέο μοντέλο το οποίο ε, ξεκινάει να εφαρμόζεται. Και επίσης τι γίνεται με τα προγράμματα πλαίσιο. Η σχέση με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο εμφανίζεται και εξαφανίζεται και δεν ξέρω πολύ καλά πώς ε, αλληλοσυνδέονται αυτά. Τώρα στη νέα χρηματοδότηση όπου ένα πολύ σημαντικό ε, τμήμα του εβδόμου προγράμματος πλαίσιο περιλαμβάνεται θα θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν πώς λειτουργούν όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα στοιχεία για τον μελλοντικό προγραμματισμό. Θέλει να παρέμβει ο εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου για τα όσα είπε η κυρία Γιάλα Σέντερ. Yes, thank you. Ναι, θα ήθελα. Να ξεκινήσω με τα σχόλια του κυρίου ότι οι λόγοι αποτυχίας ε, είναι, του κ. μάλλον, είναι η αποτυχία του ιδιωτικού τομέα. Η αγορά ουσιαστικά δεν ήταν έτοιμη για να προωθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ε, ουσιαστικά παραπλάνησε τον ε, δημόσιο τομέα. Όταν φτάσει σε μια κατάσταση ένας αγοραστής, ένας πολιτής, τα πράγματα ε, ξεφεύγουν, ε, δεν τήρησε τον προπολογισμό και τις προθεσμίες. Τι μαθήματα διδαχθήκαμε από τις δυσκολίες του προγράμματος. Καταρχάς θα πρέπει να έχουμε κάποια σημεία αναφοράς. Πρέπει να δούμε και να κινηθούμε με βάση την βιομηχανία. Σε αυτή τη διαστημική, ε, τα διαστημικά αναπτυξιακά προγράμματα ε, είχαμε παλιά σημεία αναφορά με 40% χρηματοδότηση. Επίσης, ήταν χρήσιμη η συμμετοχή του δημόσιου τομέα. Ε, όταν ανέλαβε ο κύριος Μπαρό, ουσιαστικά είχαμε φτάσει σε μια διαδικασία διάσωσης. Ήρθα σε επαφή με τον κύριο Μπαρό και νομίζω ότι συμφωνούμε με αυτά που λέει η έκθεση. Κυρία Γιάλα, το δικαστήριο ανά, ε, ανέλησε πώς απέτυχε αυτή η εταιρική σχέση δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Τώρα τι θα συμβεί στο μέλλον. Ε, μπορούν αυτές οι εταιρικέ σχέσεις ε, να κρατηθούν σε επίπεδο ανταγωνιστικό. Αν υπάρχει ανταγωνισμός και ανταγωνιστικότητα, αυτό είναι το κλειδί. Ε, αν δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ο ιδιωτικό τομέα πετάει τον μπαλάκι και τι δυσκολίε ε, στον δημόσιο τομέα. Πρέπει να ανταγωνίζεται ο ένα τον άλλον. Τώρα, τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε, το follow-up. Μετά από μια τέτοια έκθεση ε, δεν μπορεί να υπάρξει follow-up ούτε για το Γαλιλαίο ούτε για τις άλλες κοινέ επιχειρήσεις. Τώρα για τον προϋπολογισμό δεν είναι θέμα μόνο του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά και θέμα των ανθρώπων που παίρνουν τι αποφάσει. Εμείς θα κανονίσουμε πώς θα κινηθούμε σε περίπτωση που έχουμε πολιετή προγραμματισμό και ξεπερνάμε τι χρηματοδοτικέ προοπτικέ. Θα συμφωνήσουμε πώς θα συνεχίσουμε, πώς θα κάνουμε κάποιες προβλέψεις. 10 ε, με 40% είναι τα πρότυπα της βιομηχανίας. Οτιδήποτε άλλο θεωρείται αποτυχία. Για τη σχέση με το, με το πρόγραμμα πλαίσιο, Το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο ήταν ουσιαστικά το πιο επιτυχημένο κομμάτι. Και νομίζω ότι εδώ η Κομισιόν και το Ελεκτικό Συνέδριο ε, συμφωνούν ότι ουσιαστικά θα υπάρξει μια θετική εξέλιξη ε, και θα διδαχθούμε από τα παθήματα. Merci, Monsieur le Président. Euh, je suis Bonucci euh, de la DG από τη Γενική Διεύθυνση Τρέν. Καταρχάς, να συγχαρώ το Ελεκτικό Συνέδριο για την έκθεση και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την προσπάθειά του. Πρέπει να διευκρινίσουμε πριν να υπησέλθουμε σε υπερβολικές αναλύσεις για τα πεπραγμένα του παρελθόντος. Πρέπει να πούμε λοιπόν το πλαίσιο σήμερα άλλαξε άρδιν. Η Κομισιόν ε, στο τέλος του 2006 είχε ήδη ενημερώσει για τις δυσκολίες που η εταιρική αυτή σχέση είχε αντιμετωπίσει και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος είχε μιλήσει για τις τεχνικές δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει αυτά τα σύνθετα και εντελώς καινοτόμα προγράμματα. Σήμερα η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η απόφαση να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της Κομισιόν μας έδωσε έναν ηγετικό ρόλο εμάς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τελείως διαφορετικό από το όλο που παίζαμε ε, στην περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Δηλαδή, από τον Απρίλιο του 2009 ανακτήσαμε την πλήρη ευθύνη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Δηλαδή φέτος, στους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ενεργητικά στοιχεία της ε, υπηρεσίας θα τεθούν, θα μπουν στον προϋπολογισμό θα καταγραφούν. Επομένως, μια απάντηση στο ποιος είναι ιδιοκτήτης πιανού πράγματος. Σε ό,τι αφορά τώρα το Γαλιλαίο, όπως προβλέπει και ο κανονισμός, περάσαμε, έχουμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος που καθορίζει τον ε, ρόλο των μεν και των δε. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια μορφή διαχείρισης τελείως διαφορετική από αυτή που είχαμε το 2005-2006. Τρίτον, Α πάμε στα ουσιαστικά στοιχεία της ε, σύσταση του δικαστηρίου, του ελεκτικού συνεδρίου, συγγνώμη. Δεν είχαμε το απαραίτητο προσωπικό τότε, το 2005-2006, για την αποτελεσματική διαχείριση. Τώρα έχουμε κάποιους ε, εμπειρογνώμονε και αυξήσαμε το συνολικό προσωπικό που ασχολείται με το πρόγραμμα Γαλιλαίος, ε, μέσα σε κάποια εύλογα πλαίσια βέβαια. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε 75 με 85 άτομα που δουλεύουν 100% ε, πάνω στο Γαλιλαίο. Τώρα, ο ρόλος με τους εταίρους ε, και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος επανακαθορίστηκαν. Και ο διαθεσμικός χαρακτήρας έχει εξασφαλιστεί χάρη σε μια ομάδα διαθεσμική που συνεδριάζει περιοδικά για να δει που βρίσκονται τα πράγματα. Αυτά για τη διαχείριση τη σημερινή. Τώρα, ποια είναι η θεώρησή μα, το όραμά μα για το Γαλιλαίο. Εμείς δεσμευτήκαμε για να δώσουμε μια έκθεση στι αρχέ του 2010 στο Κοινοβούλιο που θα εξηγεί τα πράγματα και που θα προτείνει διάφορες εναλλακτικέ λύσεις. Θα, με βάση τους στόχους και πώς θα περάσουμε από μια φάση σήμερα που είναι φάση υλοποίησης σε μια φάση εκμετάλλευσης. Είμαστε σε φάση προετοιμασία ακόμα και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια θα άρει κάποιε από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου και του εισηγητή. Ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ. Ε, ε, καλύφθηκα από, την, από τα σχόλια που έγιναν το Ελεκτικό Συνέδριο και την Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος ε, Γκέρμπραντι. Ευχαριστώ και το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον ε, εισηγητή κύριο Λιμπεράτσκι για την ε, αξιόλογη συμβολή τους και για τις πολύ σαφείς εισηγήσεις τους, ειδικά από τον εισηγητή, τον κύριο Λιμπεράτσκι. Εάν αναλογιστούμε το στρατηγικό ενδιαφέρον του προγράμματος αυτό για την Ευρώπη, τα γεγονότα είναι εντυπωσιακά, διότι χάθηκε τελείως ο έλεγχος της διαχείρισης, αμφισβητήθηκε ο ρόλος των κρατών μελών και διάφορα άλλα δεινά. Τώρα, όπως είπε ο κύριος Λιμπεράτσκι, η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου λέει ότι το κάθε κράτος μέλος προασπίστηκε τα δικά του τα συμφέροντα και προσπάθησε να προαγάγει τα συμφέροντα του δικού του βιομηχανικού τομέα, γεγονότα τα οποία δεν είναι διόλου ανθαρρυντικά για το πρόγραμμα αυτό. Και πάρα πολλοί άλλοι φορείς ήταν επικριτικοί κατά του Γαλιλαίου, παρόλο το μεγάλο στρατηγικό ενδιαφέρον που έχει και η δική μου κυβέρνηση και το, ο Υπουργό Οικονομικών εξ αρχής είχε πει ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα η ύπαρξη του προγράμματος Γαλιλαίου. Είχαν λοιπόν πολλά κράτη-μέλη απολύτως αρνητική στάση και αυτή η άρνηση συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση την τεράστια του κόστους, στις μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν. Υπάρχει πράγματι ε, υπήρχε εξ αρχής μεγάλη ανησυχία για το κόστος και τελικά οι προφήτες αυτή τη της καταστροφής ε, αποδείχθηκαν σωστοί. Το κόστος ξέφυγε ελέγχου ε, και, σε αυτό βοήθησε και η πολύ μπερδεμένη και συγκεχημένη δομή διαχείρισης, management. Grazie. Se vuole prendere la parola la Commissione sul το λόγο για το ερώτημα που έκανε ο βουλευτής. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο που έχουμε σήμερα νομίζω ότι μας επιτρέπει να τελεσφορήσουν τα προγράμματα μέσα στις προθεσμίες που έχουν καθοριστεί με βάση τις τεχνικές δυσκολίες. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο πρόγραμμα και δυνάμει της ε, ταχύτητας που μας, που μας επιτρέπουν τα δεδομένα. Όπως παράδειγμα το χάρη το procurement. Με βάση τα όσα κάναμε το 2009 και εξαλθούμε να κάνουμε, το νέο χρονοδιάγραμμα που αποφασίστηκε βάσει του κανονισμού, του νέου κανονισμού, Νομίζω ότι σεβόμαστε πλήρως του τους στόχους και θα υλοποιήσουμε πλήρω του στόχου που έχουμε θέσει. Άλλο κανεί. Ευχαριστώ όλου του εκπροσώπους τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ελεκτικού Συνεδρίου για την συνεισφορά του στην εποφελή συζήτηση. Να υπενθυμίσω τις επόμενες ε, συνεδριάσεις 3 Νοεμβρίου και 4 Νοεμβρίου και 10 Νοεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, κλείνει η συνεδρία και θα τα ξαναπούμε στις 3 Νοεμβρίου. Α, Alt. Η κυρία Αντρεάσεν. Yes, I would like to demand... Uh, θα ήθελα να ζητήσω μία αλλαγή στα πρακτικά της 26ης, 21ης Ιουλίου. Θα ήθελα να περιληφθούν όλα τα ονόματα των Ευρωβουλευτών που ψήφισαν την, ε, για την αντιπροεδρία αυτής της Επιτροπής, πρακτικά 21η Ιουλίου. Θέλει κανείς το λόγο για το θέμα αυτό. Κανένας. Ωραία. Por favor, es que no sé muy bien lo que να ρωτήσω αν μπορούμε να ζητήσουμε ονομαστική πληροφορία κατόπιν Δεν κατάλαβα τι μα ρώτησε η κυρία Αντρέασεν, διότι το σημείο της ε, προεδρίας των, ε, της, συγγνώμη, των αντιπρόεδρων είναι πολύ σαφέ. Ε, τι θέλετε να γράψουμε ονομαστική ψηφοφορία ε, δεν κατάλαβα τι ακριβώς ζήτησε η κυρία Αντρέσεν. Ε, εμείς έχουμε το δικαίωμα να το γνωρίζουμε. Μπορεί να μην κατάλαβα καλά. Τι ζητάτε. κύριε Αντρέσεν, παρακαλώ, θέλετε να διευκρινίσετε. Ζητάω όχι να αναγράψετε ονομαστικά τα άτομα. Θα ήθελα τα ονόματα των ανθρώπων που ψήφισαν να συμπεριληφθούν κατα... Ε, στα πρακτικά. Είτε υπέρ είτε κατά. Δεν ζητάω να ε, γράψετε τι ψήφισαν, αλλά τα ονόματα αυτών που ψήφισαν. Και ο λόγος που το ζητάω είναι διότι εξαφανίστηκε αυτό το κομμάτι της ε, συνεδρίασης. Με καταψήφισε η Επιτροπή ως υποψήφια αντιπρόεδρο και εξαφανίστηκε αυτό το κομμάτι στα πρακτικά. Άκουσα αυτά που είπατε. Πραγματικά εκπλήσωμαι όμως. Ουσιαστικά αυτό που λέτε είναι απόπειρα λογοκρισίας. Εμείς έχουμε κατάλογο συμμετοχόντων στην Επιτροπή. Δεν είναι μυστικό. Είναι ένας κατάλογος ο οποίος είναι διαθέσιμος και είναι στη διάθεση σε όλα τα πρακτικά δεν υπάρχει καν υποχρέωση ψήφου, υπάρχει δικαίωμα ψήφου και ο κατάλογος των ε, παρόντων ουσιαστικά υποδεικνύει ποιο απολάβανε αυτό το δικαιώματο εκείνη την ημέρα. Και νομίζω το θέμα πρέπει να θεωρηθεί λήξαν εδώ. Παρακαλώ, κύριε Ανδρέασεν. Δεν πιστεύω θέμα. Δεν έχει τελειώσει εδώ το θέμα, γιατί ο κατάλογος των ε, συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερο από τον ε, κατάλογο των ανθρώπων που ψήφισαν. Ευχαριστώ. Αυτό συμβαίνει διότι δεν ψήφισαν όλοι οι παρόντες. Εγώ έχω το δικαίωμα και είναι προνόμιο μου να ψηφίσω, αν όμως θέλω, δεν είμαι υποχρεωμένος να ψηφίζω. Γι' αυτό ακριβώς η λίστα των παρόντων φτάνει και περισσεύει και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και όσοι θέλουν ψήφισαν. Eh, Επιμένει η κυρία Αντρεάσεν, μπορούμε να ψηφίσουμε. Μια και είναι έτοιμα βουλευτού, μπορούμε να αποφασίσουμε. Ψηφίζοντα. Ποιο είναι υπέρ, ποιο είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ του αιτήματο τη κυρία Αντρεάσεν. Να σηκώσει το χέρι, παρακαλώ. Και Ποιος είναι κατά. Απορρίπτεται το αίτημα. 5-4. Γεια σας. Πρέγω. Γράψε στα πρακτικά ότι το ζήτησα και απορρίφθηκε. Ζήτησε αυτόν τον κατάλογο και απορρίφθηκε. Βεβαίω και θα το γράψουμε, λέει ο Πρόεδρος. Πρέγω. Sí. Yo, yo también le pediría al secretariado que nos... Θα ήθελα να ζητήσω από τη Γραμματεία να μας πει εάν ε, επιτρέπεται από τον κανονισμό αυτό το αίτημα. Ο κύριος Λιντεράσκη το είπε, υπάρχουν τα πρακτικά και γράφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Εάν δεν υπήρχε προηγούμενο αίτημα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Ποτέ δεν τίθεται τέτοιο θέμα, εκτός και αν ζητάμε αν υπάρχει απαρτία, που είναι το μόνο ερώτημα που κάνουμε, ή ονομαστική ψηφοφορία. Έτσι εκ των υστέρων δεν ε, ξέρω αν ισχύει, θα ήθελα να μου πει η γραμματεία αν εφαρμόζουμε τον κανονισμό ή αν καινοτομούμε. Μπορεί να είναι καλό, αλλά θα ήθελα ήθελα να ξέρω εάν είμαστε εντός του κανονισμού, γιατί είναι πρώτη φορά που υπάρχει τέτοιο αίτημα.